Okay, colleagues, we did give people a bit more time, given that. Um, Παρακαλώ, συνάδελφοι, θα δώσαμε λίγο χρόνο γιατί ξεκινάμε νωρίτερα από ό,τι συνήθω, Από ό,τι μόλι μου είπανε, αυτό θα γίνει ε, πάγια πρακτική από εδώ και πέρα για την Τρίτη και την Τετάρτη, γιατί ξέρω ότι οι συνάδελφοι οργανώνουν και άλλε συνεδριάσει το μεσημέρι. Και εγώ μάλιστα είχα και τον Καναδό πρέσβη και χρειάστηκε να ε, διεκπαιρεώσω στα γρήγορα τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 14. Η υποβολή της έκθεσης στην Επιτροπή από την επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, του ΙΚΟΣΟΚ ε, των Ηνωμένων Εθνών που είναι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είχαμε μία αντιπροσωπεία στην οποία επικεφαλής θα ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό λοιπόν. Έχουμε δύο μέλη της αντιπροσωπείας. Μπορούμε να σας πούμε τι κάναμε, αλλά και το τι θα κάνουμε στη συνέχεια για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Νελ Δέβα, ο Μπόγκταν Βέντα, η Ανελίζε, η Χάιντι Χάτολα και οι υποφαινόμενοι πήγαμε. Και τι γίνεται. Κάθε χρόνο τα Ηνωμένα Έθνη οργανώνουν έναν πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου και ε, από εδώ και πέρα θα γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο, θα γίνεται ένας απολογισμός του που βρισκόμαστε με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει δύο τμήματα η όλη διαδικασία. Υπάρχει μια θεματική πλευρά όπου συζητιούν ε, τα διάφορες θεματικές ενότητες, ε, τα συμβαλόμενα μέρη και το δεύτερο τμήμα είναι μια συνολική αναθεώρηση. Για φέτος ε, τα θέματα ήταν ο στόχος 1 που είναι η ένδυα, ο στόχος 2 ε, μηδενική πείνα, στόχος 3 υγεία, 5 φύλλο, 9 που είναι αξιοπρεπής εργασία. Δεν μπορώ να διαβάσω καν τις σημειώσεις μου. Ε, ξέρω αυτά που αναθεωρήσαμε, αλλά δεν τα θυμάμαι απ' έξω φυσικά τους στόχους, ποιος αριθμός είναι ο κανένας. Και έχουμε και το στόχο 14 ή ε, ωκεανοί. Και κάθε χρόνο θα αναθεωρείται ο στόχος 17 που είναι η εταιρική σχέση και αφορά κυρίως τα χρήματα. Ε, ο στόχος 17 είναι κατά πόσον εφαρμόζονται ε, όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο. Τι γίνεται, έχουμε μια συνεδρία σε δύο εβδομάδων. Η εβδομάδα αυτή ήταν η θεματική ενότητα η πρώτη εβδομάδα. Εμείς δεν ήμασταν εκεί, αλλά πήγαμε στη δεύτερη εβδομάδα που ήταν οι διμερεί σχέσει, που τα κράτη-μέλη ανέφεραν τι ε, έχουν επιτύχει αυτά όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμη ανάπτυξη. 43 χώρες υπέβαλαν εκθέσει, μεταξύ ε, των οποίων και 10 ε, ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω χώρο, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σουηδία. 10 χώρες. Πέρσι η Εστονία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Φιλανδία επέβαλαν εκθέσεις. Μέχρι τώρα δηλαδή τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, υποβάλει έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Το απογοητευτικό αυτών των ετήσιων εκθέσεων ήταν ότι κάποια κράτη-μέλη επέλεξαν κάποιους συγκεκριμένου στόχους τους οποίους θα θέλουν να επικεντρωθούν, διαλέγουν δηλαδή και αυτό έχουμε πει ότι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και κάποια κράτη-μέλη δεν δίνουν το καλό παράδειγμα και δεν υπάρχει και συνέπεια μεταξύ των εκθέσεων. Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν την έκθεση που θέλουν, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο ώστε να γίνεται η έκθεση με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα πούν αν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, απλώ να κάνει κάποιο αντί να κάνει μια αυθαίρετη έκθεση, ε, δεν έχουμε συζητήσει, για παράδειγμα, στα άτυπα συμβούλια για το πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κάνουν εκθέσεις ε, στο ε, φόρουμ αυτό. Ε, εάν λοιπόν μπορούμε να είναι μια πρόθεση αυτό, να προσπαθήσουμε να συντονιζόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί ακόμα και οι εκθέσεις από τα κράτη-μέλη που είναι συγκρίσιμες δεν μπορούν να μας δείξουν εύκολα τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Έγιναν και κάποιες συναντήσεις, συναντήσαμε τον νέο επικεφαλής του UNDP, τον Ακίμ Στάινερ, το νέο αναπληρωτή Γενικό Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, τον Αμίνα Μοχάμετ, ο οποίος ε, πριν εργαζόταν στην κλιματική αλλαγή, στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Η Αμίνα Μοχάμετ είναι υπεύθυνη για την ε, εποπτεία και συντονισμό του νέου συστήματος ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα γίνει μεγάλη μεταρρύθμιση και η Αμίνα εποπτεύει όλη αυτή την αλλαγή. Και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικέ οι συναντήσει και με τον Ακίμ Στάινερ και με την Αμίνα Μοχάμεντ. Ιδίω η Αμίνα Μοχάμεντ επικεντρώθηκε ε, στην πράξη, με πρακτικό τρόπο πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που θέλουμε και μας ρώτησε συγκεκριμένα εάν ε, συνεργαζόμαστε και με τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά κοινοβούλια άλλων χωρών. Είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι χώρε να κάνουν κτήμα του αυτού του στόχου και να προσπαθήσουν να προωθήσουν τα θέματα και σε άλλε χώρε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και πρέπει να σκεφτούμε εδώ πώ ε, μπορούμε να προωθήσουμε αυτού του στόχου. Αναφέρθηκε επίσης και στην ΑΕΤ ως χώρα ε, την οποία θα μπορούσαμε να προσέξουμε και την Ιγυρία που είναι δική της η χώρα. Έχουμε και κάποιες γυναίκες από την Ιγυρία εδώ σήμερα και καλό είναι να το δούμε και αυτό. Συναντηθήκαμε επίσης με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ταμείου Πληθυσμών των Ηνωμένων Εθνών, την Νατάλια Κάνεμ, η οποία αναφέρθηκε ε, στα όσα έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, ε, τη, ε, ε, πρόβλημα υπάρχει με τη χρηματοδότηση για τον οικογενειακό προγραμματισμό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και όπως ξέρουμε τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να προχωρήσουν το θέμα αυτό στα θέματα γυναικών για να υπάρξει στήριξη για τις γυναίκες ε, μέσω της δικής της χρηματοδότησης. Συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον Άντο πρόεδρο, συγγνώμη, Μαχμούντ Μοχελτίν και τον ε, ειδικό εκπρόσωπο για τη Διεθνή Μετανάστευση των Ηνωμένων Εθνών, τη Λουίζα Άρμπορ και η Λουίζ Άρμπορ είναι ο νέος σύνδεσμος των ΟΕΕ για τη μετανάστευση. Ήταν δικηγόρος για διεθνή δικαιώματα. Νομίζω ότι ήταν εισαγγελέα σε υποθέσεις ε, στο ε, δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ήταν εντυπωσιακή. Είναι Καναδί και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επικεντρώνονται ε, στα νομικά μέσα στη μετανάστευση στον Καναδά, να απομακρύνουν αμέσως τους ανθρώπους από την κατάσταση του πρόσφυγα δηλαδή. Και νομίζω ότι μπορούμε να διδαχθούμε πάρα πολλά από τις άλλες χώρες και επίσης ε, μάθαμε και λίγα περισσότερα για το πώς θα λειτουργήσει το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση. Ήταν και άλλοι συνάδελφοι εκεί, δεν θα μιλήσω εξ ονόματό του. Ξέρω ότι μία συνεδρίαση που πήγαμε ήταν πολύ χρήσιμη και καλό θα ήταν να έχει η Επιτροπή μα μία εικόνα για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη με του στόχου ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ω Επιτροπή δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και επίση είχαμε το δίκτυο βιώσιμη ανάπτυξη και το Ίδρυμα Bertelsmann που μα παρουσίασαν την έκθεση του 2017 για του δείκτε των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη πώς προχωράμε για τα διάφορα θέματα, πώς προχωράει κάθε χώρα. Και η ιδέα ήταν να τους προσκαλέσουμε και σε μια μελλοντική συνεδρίαση. Μια άλλη ιδέα θα ήταν, επειδή ε, έχουμε τον Νοέμβριο τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπου προσκαλούμε και τις ε, Επιτροπές ε, Διεθνούς Ανάπτυξης από τα διάφορα Εθνικά Κοινοβούλια, καλό θα ήταν να ξέρουν και τι υπέβαλαν οι χώρες τους στα Ηνωμένα Έθνη και να γίνει μια σύγκριση μεταξύ αυτών. Γιατί δεν θα πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης εάν δεν πιέσουμε και εμείς τις κυβερνήσεις μας ε, να πιέσουν ε, τα θέματα αυτά στις χώρες τους. Ε, συναντηθήκαμε επίσης και με μέλη της Κόγκορτ, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να πω ε, από πλευρά μου ευχαριστώ πολύ στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη που ήταν εξαιρετική, μας στήριξε με εξαιρετικό τρόπο και κυρίως την Κάθριν, δυστυχώς δεν θυμάμαι το επιθετό της, αλλά ήταν πάρα πολύ ε, εξυπηρετική. Κάθριν ας! Χες, δεν μπορώ να το προφέρω, ο Κριστιαν θα πρέπει να σας το πει ή να μην το γράψει για να μπορέσω να το προφέρω. Είναι πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη που μας προσέφεραν και αυτή και ο πρέσβης και το προσωπικό και η Επιτροπή Επιτόπου. Επομένως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στους υπολείπους. Ε, ε, θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης πλέον και νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε γι' αυτό. Γιατί του χρόνου ε, θα συναντηθεί και πάλι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου. Το 2019 τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει έκθεση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολη η στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα είναι και αμέσω μετά τι εκλογέ. Ε, Αυτή που θα είναι ακόμα εδώ, η Γραμματεία για παράδειγμα, ε, μπορούν εντωμεταξύ να προετοιμαστούν με τις αντιπροσωπείες ε, της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, της νέας Επιτροπής Ανάπτυξης, για να πάνε στο πολιτικό φόρουμ τον Ιούλιο του 2019. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να πάμε εκεί ως αντιπροσωπεία, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει έκθεση για τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς θα γίνει δεν ξέρω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε αντιπροσωπεία και να υπάρξει αυτόματα. Θα είναι η εβδομάδα αμέσως μετά τη συγκρότηση των νέων ε, επιτροπών. Θα υπάρχει πρόεδρος επιτροπή στο μεταξύ. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται, αλλά ε, σίγουρα η Επιτροπή μας θα βοηθήσει να προετοιμαστεί η ε, αντιπροσωπεία αυτή, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Βλέπω κάποιους από τους συναδέλφους που ήταν εκεί, δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως σας είπα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό μας που διοργάνωσε αυτή την εξαιρετική επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και ε, είχε μεγάλη σημασία να αντιπροσωπεύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ήμασταν ε, επιτυχής στο να ε, μεταδώσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας. Και ε, θέλαμε κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής να λάβουμε υπόψη αυτή τη μεταρρύθμιση που, στην οποία θέλει να προβεί ο νέος Γενικός Γραμματέας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται αυτές οι αλλαγές με βάση τα παγκόσμια συμφραζόμενα και χαίρομαι διότι αυτό αποτελεί μέρος και της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε επικεφαλής αυτού του νέου οικοδομήματος. Τα ζητήματα τα οποία θίξαμε και στην Ευρώπη είναι τα ίδια, δηλαδή στόχοι βιώσιμης χιλιετίας, ο ιδιωτικός τομέας, η ασφάλεια, η ειρήνη και η μετανάστευση και αυτή η συνάντηση με τον κύριο Άρμπορ είχε πολύ μεγάλη σημασία διότι ασχοληθήκαμε με θέματα μετανάστευσης. Πρόκειται για παγκόσμιες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα με όλους τους εταίρους. Και φυσικά εγώ, ο Νόρμπερτ και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη συνένεση. Τέλος, ε, θεωρώ ότι με αυτή τη συνάντηση η Επιτροπή θα εφαρμόσει πολύ καλύτερα τους ε, στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης για το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εποπτεία και λογοδοσία. Και Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και μία περαιτέρω συνάντηση για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. αυτό που έχει σημασία είναι και η συνεισφορά μας και ε, το, το γεγονός ότι έχουν επιπτώσει αυτοί οι στόχοι και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είδαμε τι γίνεται στην ε, Καραϊβική, στον Άγιο Μαρτίνο και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Τα είδαμε αυτά με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα τα οποία δεν προελέχθησαν. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση στο Ηνωμένο, στα Ηνωμένα Έθνη και η Δανία και η Εστονία ασχολήθηκαν με θέματα διατροφικής αλυσίδας και είδαμε πώς οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης εντάσσονται στους γενικότερους στόχους και αυτό ε, αφορά και τη νέα πρωτοβουλία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και είδαμε πώς η Ιδανία και η Εσθονία ασχολούνται με τον τομέα του επιχειρήν και αυτό αφορά και το φόρουμ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις όλο και αναπτύσσονται και προωθούν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει διάλογος όλων των χωρών, γιατί δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγω όλες τις χώρες ή όλες οι χώρες. Γι' αυτό υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Και όπως ξέρετε, η Γερμανική Οργάνωση Χημικών προβλέπει μία συνεδρίαση τον Δεκέμβριο για την διατροφική αλυσίδα και την χρήση χημικών ουσιών μέσα στα πλαίσια των στόχων. Και στις 21 Νοεμβρίου θα έχουμε τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, την ε, διακοινοβουλευτική συνάντηση και εδώ θα μπορούσαμε να δούμε ποιες είναι οι μέχρι του δε εξελίξεις. Και υπάρχει και με στα πλαίσια της Περιφερειακής Επιτροπής η SDG Watch και άλλες οργανώσεις που συμμετέχουν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και πέρα από αυτό, έχουμε και το θέμα της επεξήγησης των μηχανισμών για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί σε εθνικό επίπεδο. Ο Τίμερμανς και η Μογκερίνη ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα ήδη από το 2015 όταν παρευρέθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ο Τίμερμανς δεν μου απάντησε στην πολιτική μου ομάδα σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ως προς τους στόχους. Γιατί έχουμε την κυκλική οικονομία και άλλα ζητήματα τα οποία συμβαδίζουν αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν από πλευράς στόχων. Πέρα από αυτό είχαμε και ένα μέλος από την Επιτροπή Προϋπολογισμών που μας μίλησε για τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας καθώς και ο έλεγχος του προϋπολογισμού για την ε, πλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και από πλευράς προϋπολογισμού και θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τους ε, στόχους του πολιετούς πλαισίου έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου να ανταποκριθούμε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους της Νέας Υόρκης. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στην Επιτροπή ότι το MFF είναι βασικό μέσον για την πλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ε, Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι σοσιαλιστές έχουμε προωθήσει και ένα έγγραφο σε σχέση με την αναπτυξιακή ε, πορεία της Αφρικής και υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα σε επίπεδο ε, fellows για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε και το σχέδιο GSZ. Γιατί όταν, ρωτήσαμε την, όταν ρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, δεν μπορούσε να γνωρίζει ακριβώς πώς είχε συγκεφαλαιωθεί η κατάσταση για να ξέρουμε πόσο έχουμε προχωρήσει σε επίπεδο GSZ. Όμως το προσωπικό της Νέας, από τη Νέα Υόρκη μας υποστήριξε και από πλευράς Παγκόσμιας Τράπεζας πέρα από τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό στην επόμενη συνάντηση η Ευρωπαϊκή Επίτροπη θα πρέπει να είναι παρούσα, δηλαδή η ομάδα του Τίμερμανς που ασχολείται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η νέα συνάντηση θα γίνει το 2019. Ευχαριστώ πολύ. Γκέρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ανησυχεί ιδιαίτερα η βραδύτητα χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και θα ήθελα η Επιτροπή που είναι παρούσα σε όλες μας τις συνεδριάσεις να μας κάνει μια πρώτη ένα πρώτο απολογισμό του τρόπου με τον οποίο η ίδια αλλά και τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρώτο. Δεύτερο και σχετικό με το προηγούμενο, οι μεθοδολογίες που υλοποιούνται για την ε, αξιολόγηση των ε, μεθόδων είναι ευρωπαϊκή μεθοδολογία ή πηγαίνει κράτος προς κράτος. Γίνεται μια διάγνωση των εξελίξεων ανακράτος, τονίζονται τα σημεία που υπολείπονται ιδιαίτερως, πώς θα προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει περισσότερη προσπάθεια συντονισμού από πλευράς των ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό που ανησυχεί εμένα είναι ότι μας απασχολεί η θέση ε, σε εφαρμογή αυτών των μηχανισμών, ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα τρόποι μέτρησης πάντα μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης, αλλά με ποια μέθοδο θα υλοποιείται αυτό. Και τελευταία παρατήρηση. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε την ανάγνωση των ε, πραγματοποιηθήσεων προόδων κράτος προς κράτος. Αλλά η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο που έχει συνέπειες για όλα τα κράτη-μέλη και το έχουμε πει πολλές φορές σχηματικά, εγώ προσωπικά το έχω υπενθυμίσει πολλές φορές εδώ, η παγκοσμιοποίηση γεννά πλούτο, ανάπτυξη χρόνο το χρόνο, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση πάνω από το μέσο όρο των οικονομικών μεγεθών στα κράτη που έχουν μέσα μεσαία ανάπτυξη, μεσαίο επίπεδο αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και τις ανισότητες μέσα σε κάθε κράτος. Άρα υπάρχει ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο δηλαδή, που φέρνει τα αποτελέσματα που σας εξηγώ σε εθνικό επίπεδο, ως παγκόσμιο επίπεδο λοιπόν η παγκοσμιοποίηση, μπορεί να φέρνει ανισότητες μέσα σε κάθε κράτος χωριστά. Τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πλούσια αλλά και τα φτωχά κράτη, τα κράτη με μεσαίο εισόδημα όσο και τα πλούσια κράτη μπορεί να έχουν διαφορετικές ε, συνέπειες από την παντοσμοποίηση. Αυτό δεν το καταγράφουμε και αυτό που ρωτώ είναι εάν υπάρχουν κάποιες πραγματικές απόπειρες επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, επί για να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα δώσει απαντήσεις ή θα μας επιτρέψει να αντιδράσουμε κατά τρόπο οικουμενικό σε ένα οικουμενικό πρόβλημα. Γιατί το να αντιδρά ο καθένα με τα εθνικά του μέσα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα. Σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα που πρέπει να μα απασχολήσει. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει η Επιτροπή να μα δώσει κάποιε απαντήσει και για να τελειώσω έχω αποστείλει στην κυρία Μέρκελ επιστολή όταν, ήταν, ε, όταν είχε την προεδρία του G20 για να τις εκθέσω το πρόβλημα αυτό. Με μια συγκεκριμένη πρόταση στην επιστολή μου. Να καταγραφεί μια προσέγγιση όπως αυτή απαιτείται για την ε, αξιολόγηση της υφόρου ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέσα από το G20 γιατί διαφορετική είναι η μελέτη του ζητήματος στα Ηνωμένα Έθνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη-μέλη ή στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει ένας χώρος συζήτησης ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και είναι απογοητευτική η πολιτική η οποία υλοποιείται, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ένας ενιαίος χώρος ο οποίος θα είναι και αποδεκτός και θα επιτρέπει την πρόοδο. Μου απήντησε ο κύριος Αλτμαερ, υπουργός ε, προεδρίας, καγκελαρίας δηλαδή, μου είπε ότι α, καθυστέρησε η επιστολή σας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εάν αυτό είναι η απάντηση, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε για μια προσεχή συνεδρίαση του G20. Και είναι απαραίτητο όλες οι αρχές και κυρίως εκείνες οι οποίες ε, είναι και προσφορότερες για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων να στηριχθούν με κάθε μέσον, με την πυθό ή αν χρειαστεί και με την αμφισβήτηση, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Η Πρόεδρος Νέσαρλ, ναι, όπως είπες και εσύ, όταν είχαμε το, τη Σύνοδο Κορυφής και ιδιαίτερο χαίρομαι γιατί αναφέρεται στο ε, σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων η έκθεση του κύριου Πόγκα που είχαμε και χθε και σήμερα να ψηφίσουμε ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει αυτό η στόχοι της χιλιετίας, η στοχή της βιώσιμης ανάπτυξης να ε, μπουν στο επίκεντρο των συνομιλιών μας. Δεν μπορούμε περιστασιακά μόνο να τους αναφέρουμε. Πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό και όπου αλλού δει. Ε, θέλεις κάτι να πεις? ο, προ... ο κύριος Γκέρενς, ο Μωρίς Πόγκα νομίζω θέλει και εκείνος να ακούσει τη στρατηγική της Επιτροπής όσο και εγώ. Έτσι δεν είναι Μωρίς. Η Πρόεδρος. Άννη. Μια πολύ γρήγορη απάντηση. Χρειάζεται βεβαίως να συζητηθεί πληρέστερα μια παγκόσμια απάντηση θα μπορούσε παραδείγματι να είναι κάτι σαν αυτό που έχουμε στο χώρο της κλωστοϊφαντουργίας, το πρόγραμμα ECT, το οποίο επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ισότητα φύλων, μείωση των διαφορών κτλ. Κάτι που μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Και έχουμε μια αρχική έκθεση για την διπλωματία παραδείγματι τη σχετική με την κλιματική αλλαγή εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια λύση. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε στην Επιτροπή μας, από την Επιτροπή μας το θέμα των βιώσιμων στόχων, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, να μπει στην ε, ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν τρόπο τακτικό, πρακτικό και το πολιτικό μας έργο θα πρέπει να είναι ακριβώς να εξηγούμε την πολιτική μας στρατηγική και να εξηγούμε ότι χρειάζεται να εξηγείται κάθε φορά γιατί επιδιώκονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς οι πολιτική πρέπει να το αναφέρουμε, διαφορετικά δεν το αναφέρει κανείς. Εάν δεν φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα το κάνει κανείς. Ίσως κάθε επιτροπή θα έπρεπε να αναλάβει μια έκθεση Φερρυπίν στην οποία θα τονιζόταν η υλοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ή πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε τομέα πολιτικής. Εσείς, Χάρλα, αναφέρθηκε στο G20. Έχουμε και διακοινοβουλευτική διάσκεψη εκεί. Ίσως κάποιον από το Συμβούλιο ή από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στο G20 θα μπορούσαμε να καλέσουμε κάποιον να μιλήσουμε. Ήταν η πρεπει να ενσωματωθουν σε καθε τομεα πολιτικης εσυ αλλα αναφερθηκε στο g μεγάλη διάσκεψη όπου ε, έγιναν ε, οι αναφορές στους στόχους αυτούς, αλλά πέραν της Μέρκελ οι Γερμανοί πολιτικοί δεν φαίνεται να τους έχουν εστερνιστεί. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να στήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Επιτροπή. Πολλά τα θέματα που έχουν απευθυνθεί. Κάρλος Μπερόθ Καρθία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εύα Κοράς στη συνέχεια από την Ευρω... Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής για τις παρεμβάσεις τους και τα σχόλιά τους. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών στις θελοντικές αυτές παρουσιάσεις, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ανέκυψε στην αρχή μετά τη Σύνοδο θα διαβιβάσουμε το μήνυμα ότι όσοι συμμετέχουν ε, στην διαδικασία διαπραγμάτευσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι λέτε. Θα διαβιβάσουμε το μήνυμα στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, ε, τώρα συντονίζει την όλη παρουσίαση. Και φυσικά με το επιπλέον όφιλο ότι τώρα είναι υπό την ηγεσία του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμανς και του αντιπροέδρου Κατάινεν και επομένως ε, θα πούμε ότι υπάρχει μήνυμα από το Κοινοβούλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει περιθώριο για να βελτιώσουμε τη συνέπεια. Υπάρχουν και κάποιες ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές για να βελτιωθεί η συνέπεια, αλλά ίσως δεν έγινε παρκώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι στην πρώτη περίοδο η προτεραιότητα από πλευρά Επιτροπή ήταν για να πιέσουμε κυρίω για την έννοια τη ε, υποβολή εκθέσεων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπατε και εσεί στην παρέμβασή σα και επιβεβαιώνω ότι ο στόχος είναι να καταρτιστεί η πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης το 2019. Το 2019 επελέγει, διότι όταν έγινε διαπραγμάτευση του πολιτικού φόρουμ υψηλού επίπεδου, ε, αποφασίστηκε ότι το φόρουμ αυτό θα συναντάται σε δύο επίπεδα και κάθε τέσσερα χρόνια σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Και εκεί θέλει να προβληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι δηλαδή το 2019 και από εκεί και πέρα κάθε τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, ε, ε, να σας πω ότι το 2019 ε, θα θυμάστε ίσως ότι είναι και η ημερομηνία που συμφωνήθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για την συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή της συνένεσης της ανάπτυξης που λογικά θα γίνει και αυτή τότε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει να συνεργαστούμε και από αυτού δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω για ε, φετινά, το φετινό πολιτικό φόρουμ, πέραν των όσων είπατε κι εσείς, υπήρχαν κάποιες επιπλοκές για κάποιες πτυχές της δήλωσης. Αυτό βέβαια συμβαίνει πάντα στα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρχαν ε, κάποιες εθελοντικές ε, εθνικές εκθέσεις, θεματικές εκθέσεις και μία σημαντική εκδήλωση που έγινε στο περιθώριο ε, με την επιτυχή συμμετοχή και της κυρίας Λίντα Μακάβαν για την παρουσίαση της νένεσης για την ανάπτυξη ε, στην Ομίγυρη στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Δεν αναφέρουμε στην εκδήλωση τόσο πολύ όσον αφορά στο πόσο επίκαιρο ήταν αυτό το θέμα. Θυμάμαι τη συζήτηση στην Επιτροπή ΔΕΒΕ για την έγκριση αυτή τη συνένεση. Υπήρχαν παρεμβάσει και από εσά, ε, κυρία Πρόεδρε, και από του συνεισηγητέ για το γεγονό ότι πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Ε, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ ε, ανέφερε ότι αποσύρεται από τη συνθήκη των Παρισίων και ότι πόσο σημαντικό είναι να δείξουμε πολύ ισχυρή υποστήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή αυτών των στόχων της βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίω για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι και αυτό το οποίο αφορά η συνένεση. Και επαληθεύθηκε και όλο αυτό και είδαμε και πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση και προκλήσεις όπως η ανισότητα, η βιωσιμότητα που είναι ακριβώς τα θέματα τα οποία ε, ανακύπτουν στη νέα συνένεση. Και να πω επίσης ότι πράγματι προσπαθήσαμε να το πάμε σε όλα τα επίπεδα. Συζητάτε ενεργά και στο G20 παρεπιπτόντος. Η Κίνα και η Γερμανία έκαναν ιδιαίτερη προσπάθεια και η Γερμανία ήταν πραγματικά ε, πρωτοπόρος ε, στην παρουσίαση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και Όσον αφορά την ιδέα για πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση, με τα χαρά σα ενημερώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον συμμετέχει ενεργά στην παρέμβαση του Προέδρου Γιούγκερ. Ε, στην ε, κατάσταση της Ένωσης δεν είναι η δήλωση αλλά είναι μια σειρά από που ανέλαβε για να παραδώσει κάποια πράγματα και του χρόνου υποσχέθηκε και ένα έγγραφο προβληματισμού για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για ε, τη σειρά των εγγράφων που θα έχουμε για το μέλλον της Ευρώπης θέλουμε να έχουμε και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ως σημαντική προτεραιότητα θέλει να τα θέσει ο πρόεδρος εκεί δεν θα είναι γενικόλογο θα φροντίσουμε να δούμε τι κάνουμε και τι πρέπει να γίνει. Ε, προσβλέπουμε λοιπόν και σε όλες αυτές τις εργασίες οι οποίες ξεκινούν ε, τώρα και ανακοινώθηκαν στην ομιλία και την κατάσταση της Ένωσης του Πρόεδρου. Θα πρέπει να δούμε τώρα το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για να φροντίσουμε να συμπεριληφθεί και αυτό. Για το θέμα της μεθόδου εργασίας και το πώς θα παρακολουθούμε σίγουρα αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να παρακολουθούμε διάφορες διαδρομές. Το ένα είναι οι δείκτες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά σε μερικές εβδομάδες η Eurostat θα δημοσιεύσει ε, βάση ε, των μακροχρόνιων και πολύ συχνά πολύ επιχειρησιακών ε, δικτών που προέκυψαν από τη στρατηγική του 2020 και της βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχουμε και μια πλήρη έκθεση από τη Eurostat για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με πολύ σημαντικά ε, στοιχεία παρακολούθησης και μεθόδους. Εμείς ε, δούμε και τι αναθεώρηση πολιτικών πρέπει να γίνει, κυρίως η αναπτυξιακή πολιτική βεβαίως, όπως θα φαντάζεστε. Κοιτάμε να δούμε πώς συνδέονται αυτά με τα αποτελέσματα που έχουμε, πώς μπορούμε να παρακολουθούμε τι κάνουμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξουμε προς διάφορες κατευθύνσεις. Ε, είμαστε υπόλογοι, πρέπει να δείξουμε τι ακριβώς κάναμε, πολλό δε μάλλον γιατί στη συνένεση που αποφασίστηκε μεταξύ τα θεσμικά όργανα υποσχεθήκαμε το 2019 να παρουσιάσαμε τι έχει γίνει και τις μεθόδους εργασίες οι οποίες θα πρέπει να αντανακλώνουν και τη συνένεση και τι κάνουμε όσο πλησιάζουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά μηνύματα και εγώ από πλευρά μου θα διαβιβάσω και στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε για την όλη διαδικασία του πολιτικού Φόρουμου υψηλού επίπεδου ό,τι άκουσα σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Πότε θα παρουσιάσει την έκθεση της Eurostat. Πότε θα την δημοσιεύσει, το Νοέμβριο. Ωραία, εντάξει, θα γίνει η δημοσίευση το Νοέμβριο από τη Eurostat. Ε, έχω και την ΕΙΕΔ που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ο Σάρλ όμως θα ήθελα να υποβάλει μια ερώτηση. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική, κομβικής ε, σημασίας. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια στρατηγική μεθοδολογία. Κάτι δεν πάει καλά σε επίπεδο διακυβέρνησης. Όσον αφορά τους G20, έχουμε τέσσερα κράτη, Ιταλία, ε, ε, ε, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ειδικέ διαπραγματεύσεις μεταξύ σας και των G4, δηλαδή τις τέσσερις χώρες που προανέφερα και εάν υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ Επιτροπής και G4 μέσα στα πλαίσια των G20 πώς τις επιλύεται, δηλαδή επανερχόμαστε στο θέμα της διαιτησίας όταν υπάρχει διχογνωμία επί της ουσίας. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση. Όταν θα λάβουμε την έκθεση της Eurostat, δεν θα ήταν σκόπιμο να οργανώσουμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια επί του θέματος, έτσι ώστε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει πλήρως αυτό το ζήτημα. Είμαστε στο 17 ήδη, πολύ κοντά στο τέλος της ε, θητείας. Το 2015 ορίσαμε τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε λίγα χρόνια. Θα πρέπει να επιταχύνουμε δηλαδή τους ρυθμούς μας. Θα ήθελα η Επιτροπή μας δηλαδή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να γίνει αυτή η συζήτηση το Νοέμβριο στην Ολομέλεια, αν έχει εκδοθεί πριν η έκθεση της Eurostat. Η ΕΕ θα ήθελε κάτι να πει. Η Εύα Κοράλ. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρεθήκατε στη Νέα Υόρκη, ταξιδέψατε και υποστηρίξατε ε, αυτά τα μέτρα. Και τώρα σε σχέση με τους στόχους παρακολούθησα τη γενική συζήτηση είχαμε περίπου 100 χώρες που προέβησαν σε δηλώσεις τότε και υπήρξε μια σύγκληση απόψεων σε ε, δέσμευση υψηλού επίπεδου ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως είπαν και πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής, είδαμε μεγάλες διαφορές ως προς την προσέγγιση των χωρών για τους ε, βασικούς στόχους και την ένταξή του στους εθνικούς στόχους και αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη εργασία από τα κράτη-μέλη καθώς και τα θεσμικά όργανα. Όπως είπε και ο συνάδελφος από την Κομισιόν, Είχαμε ε, μία-δύο πολύ καλές διοργανώσεις για τη νέα συνένεση, όπου και η Επιτροπή ήταν παρούσα και μπορώ να πω ότι έγιναν ε, ουσιαστικές συζητήσεις και ζωηρές συζητήσεις πέρα από την διαδικασία της συνένεσης, δηλαδή προβλήθηκαν και πολύ επικοδομητικές ιδέες από πολλούς ομιλητές ως προς τον ε, έλεγχο αυτό, το διερευνητικό έλεγχο και όπως είπε και ο Γκασπάρ Φροντίνη από την ΤΕΦΚΟ, μας ενδιαφέρει αυτός ο διερευνητικός έλεγχος και η αποτίμηση, όπως είπε και ο Κάρλος, θα έχουμε μια κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών για την εφαρμογή της νέας αυτής συνένεσης, καθώς και μια έκθεση προόδου που θα είναι έτοιμη τον Ιούλιο του 2019. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς και την πρώτη έκθεση πρόοδου το Νοέμβριο, αλλά θα γίνουν και συζητήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη για ορισμένους δείκτες, για την εκπόνησή τους δηλαδή, ως προστοιχεία, διαθεσιμότητα και ούτω καθεξής. θα λάβω υπόψη πολύ σοβαρά τις υποδείξεις σας και θα τις διαβιβάσω στους συναδέλφους. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Αυτή η έκθεση της Eurostat. Έχω αντικρουόμενα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε με τις εσωτερικές πτυχές του στόχου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά καλύπτει όλες τις πλευρές της ΤΕΦΚΟ για να ξέρουμε κατά πόσο αφορά αυτή την Επιτροπή πρωταρχικά. Κάρλος, ευχαριστώ. Είναι μια έκθεση, πρόκειται για μια έκθεση ως προς την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η, θα είναι η πρώτη έκδοση. Μετά θα έχουμε τους στόχους 1 με 16 ως προς την εσωτερική εφαρμογή αν και υπάρχει συσχετισμός με το συνολικό reporting των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα, καθώς και την εφαρμογή των εσωτερικών στόχων. Αλλά δεν έχουμε δείκτες ακόμα. Αλλά ως προς το, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 17, εδώ υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία για την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο και ένα φάσμα συναφών ζητημάτων. Αλλά το βασικό μέσον ε, αξιολόγησης θα είναι αυτή η έκθεση όπως συμφωνήσαμε με, στην όλη διαδικασία συνένεσης. Ως προς το, τους G20 υπάρχει ένα σύστημα διαιτησίας που προϋπάρχει, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αλλά επιτρέπει να ενταχθούν οι ευρωπαϊκές θέσεις σε επίπεδο G20. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται διαιτησία εδώ. Ίσως υπάρχουν αποχρώσεις, ορισμένοι φορείς εκφράζουν την άποψή τους πιο έντονα, αλλά όλοι οι φορείς γνωρίζουν ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης συμβαδίζουν με τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αποτελούν μια ευκαιρία. Και αυτό το βλέπουμε στην πρόσφατη συνένεση γιατί μιλάμε για την ευημερία, τον πλανήτη, την ε, ειρήνη και την ευημερία. Και υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση, άρα οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολύ θετικοί για την Ευρώπη μέσα στα πλαίσια της πολυμέρειας και της βιώσιμης ανάπτυξης και εντός και εκτός της Ευρώπης και πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή ελέγχου καθώς και το έγγραφο ε, αυτής της συλλογιστικής θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Προτείνω, λέει η Πρόεδρος, να λάβουμε υπόψη και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε μία συνάντηση στις 21 ε, Νοεμβρίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν ξέρω ότι εσύ είσαι ο συντονιστής, θα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με τα εθνικά κοινοβούλια, για να ξέρουν τι συμβαίνει. Και την ανάλυση της Eurostat ως προς αυτήν θα δούμε στους συντονιστές να μιλήσουμε επί του θέματος, δηλαδή ολομέλεια ή κοινή συνάντηση επιτροπών. Κάθε χρόνο θα πρέπει να προετοιμάζουμε καλύτερα το HLPF για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, ιδιαίτερα το Μάιο, εν ώψη του Μαΐου, για τις εκθέσεις που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και άλλες ε, ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας πριν από το 2019 και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε αποστολές, να μιλάμε για τους στόχους, γιατί όπως είπε και ο Άννη, αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν άλλοι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν με συστάσεις και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους στόχους και μετά θα δει και ο συνάδελφος το θέμα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή, την ΕΙΕΔ και θα συνεργαστούμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ως προς το θέμα 15 θα πρέπει να αφήσω την ε, έδρα στο συνάδελφο γιατί εγώ πρέπει να παρευρεθώ σε μια ομάδα επισκεπτών που προέρχονται από τη δική μου περιφέρεια. Γι' αυτό σας αναθέτω την Προεδρία. Okay. <coughs> Colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριος το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης προβλέπει την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής 2017, κατανόηση και αντιμετώπιση της σχέσης μεταξύ επιστημιστικής ασφάλειας, συγκρούσεων, εκτοπισμού και μετανάστευσης. Και παρακαλώ τους ειδικού μας να έρθουν στο Προεδρείο Uh, Ξεκινώ με μερικά εισαγωγικά λόγια. 16 Οκτωβρίου. Η μέρα αυτή ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Αποφασίσαμε ότι, μια, ότι αυτή είναι μία από τις παγκόσμιες μέρες που και εμείς θα πρέπει να εορτάζουμε. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ανταλλαγές απόψεων για την κατάσταση της παγκόσμιας επιστηστικής ασφάλειας. Συζητήσεις που γίνανε στην Επιτροπή μας πολλές φορές και σε συνεργασία με άλλες επιτροπές. Σήμερα άτυπα έχουμε καλέσει μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στη συνεδρίασή μας. Καθώς ε, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό, μια που αυτή η φετινή Παγκόσμια Μέρα Διατροφής ασχολείται με την σχέση της επιστηστικής ασφάλειας με την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ασφάλεια των τροφίμων και της διατροφής. 2017 λοιπόν. Ταυτόχρονα έχουμε μια πρόσφατη έκθεση και από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα ε, Τροφίμων για τις συγκρούσεις που, είναι στο, που αποτελούν τη ρίζα των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα στη διαχείριση της παγκοσμίας ε, ανάπτυξη σε συνεργασία με την ActionAid έχουμε συζητήσει τη σχέση μεταξύ της επιστημικής ασφαλείας και της μετανάστευσης και ελπίζω ότι και αυτό το θέμα θα το καλύψουν οι ομιλητές μας. Παγκόσμια μέρα διατροφής λοιπόν. Φέτος είναι μια ευκαιρία να δούμε εκ του συνεγγύς πώς σχετίζονται η μετανάστευση, οι συγκρούσεις, οι εκτοπισμοί και η επιστηστική ασφάλεια και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστούν. Καλωσορίζω τους προσκεκλημένους, τον Αρίφ Χουσέιν, την Κριστίνα Αμαράλ και τον, την Παούλινα Πιτσότο Μολίνα. Ε, θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον δόκτωρα Αρίφ Χουσάιν, Δέκα λεπτά περίπου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, στον εορτασμό, αλλά δυστυχώς δεν έχω τόσο καλά νέα. Η πρώτη έκθεση στην οποία αναφερθήκατε για το σόφι, κατάσταση δηλαδή της ε, πιστιστικής ασφαλείας στον κόσμο, ε, μια έκθεση που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο δείχνει ότι ύστερα από 10 χρόνια μείωση του αριθμού των ε, ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα, τώρα δυστυχώς αυξάνονται τα νούμερα αυτά. Από 7,77 από 777 τώρα έχουμε 815 εκατομμύρια ανθρώπων που λιμοκτονούν. Αυτό το 815 εκατομμύρια λοιπόν κατανέμοντας εξής. 60% ζουν σε περιοχές που μαστίζονται από συγκρούσεις. Τα παιδιά, 155 εκατομμύρια, κατά 75% ζουν σε ζώνες συγκρούσεως. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, η δική μου οργάνωση, δείχνει το 2016 ότι 20% των παγκοσμίων ε, πόρων για τη διατροφή μας, για τη διατροφή που προσφέρουμε εμείς, πάει σε περιοχές, 80% ε, των πόρων που διαθέτουμε εμείς πάει σε περιοχές που μας ζώντα από συγκρούσεις. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε φυσικά φαινόμενα, ε, μπορεί να έχουμε πλημμύρες, σεισμούς, αλλά και συγκρούσεις που δείχνουν από 80 σε 108 εκατομμύρια πολίτες την αύξηση των ανθρώπων που πλήττονται σε αυτές τις περιοχές οι 13 μεγαλύτερες επιστημονικέ κρίσεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουν τεράστια ποσοστά, 10 από αυτές οφείλονται σε συγκρούσεις. Γι' αυτό στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα των συγκρούσεων, γιατί είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους, και ένας από τους λόγους για οποίους αρχίσαμε να κοιτούμε το, τη συνάφεια μεταξύ συγκρούσεων, πείνας, μετανάστευσης. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για εκτοπισμούς μιλούν για 65 εκατομμύρια εκτοπιστέντες. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την ε, έκθεσή μας του Μαρτίου του 2017 που εξετάζει την πτυχή της μετανάστευσης, αλλά επιτρέψτε μου για μερικά δευτερόλεπτα να σας εξηγήσω γιατί έγινε αυτή η έκθεση και γιατί το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Είχαμε κοιτάξει το θέμα της Συρίας το 2015. Στο τρίτο τρίμηνο του 2015 διαπιστώσαμε τεράστια άνοδο του αριθμού εκείνων που έφυγαν από τη Συρία για να φτάσουν στην Ευρώπη. Ετέθη λοιπόν το προφανέ ερώτημα. Όταν η μελέτη έχει ξεκινήσει από το 2011, όταν η σύγκρουση μάλλον στη Συρία ξεκίνησε από το 2011, γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να φύγουν από τη χώρα του αυτοί οι άνθρωποι. Για να δώσουμε απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα τη έρευνα, κάναμε το εξή. Κάναμε μια εμπειρική μελέτη, ταυτόχρονα ε, επικοινωνήσαμε και ε, διατυπώσαμε ερωτηματολόγια προς εκείνους οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα τους. Η εμπειρική μελέτη εξετάζει τα αίτια της μετανάστευσης και τα δεδομένα από 125 διαφορετικές χώρες που ξεκινούν από το 1990. Διαπιστώνουμε λοιπόν ορισμένα γεγονότα εκ των οποίων το ένα που έχει και κρίσιμη σημασία είναι ότι έμεινε κατά 3, στο 3 περίπου της 100 του παγκόσμιου πληθυσμού ε, ο αριθμός των μεταναστών. 9 από τους 10 μετανάστες από την Αφρική προτιμούν να μείνουν στην Αφρικανική Ήπειρο. 8 από τους 10 Ασιάτες μετανάστες προτιμούν να παραμένουν στην Ασιατική Ήπειρο. 9 στους 10 μετανάστες που φεύγουν από τις αιστείες τους μένουν σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Κάτι άλλο, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι κάθε ποσοστό αύξησης της πείνας οδηγεί σε 2% αύξηση της μετανάστευσης. Για ένα επιπλέον χρόνο σύγκρουσης 0,4% περισσότερη μετανάστευση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο. Όταν υπάρχουν συγκρούσεις και αντίστοιχα προβλήματα, η απόφαση που παίρνει κανείς ε, ε, εκ πρώτης όψεως δεν είναι να εγκαταλείψει τη χώρα του. Υπάρχουν άνθρωποι που ε, εσωτερικά εκτοπίστηκαν στη Συρία 3, 4, 5, 6 φορές πριν φτάσουν στο Λίβανο, την Ιορδανία ή άλλη χώρα. Κοιτάω το χρόνο μου και ξέρω ότι έχω μόνο δεκαετά. λεπτά. Οι συστάσεις μας τώρα λοιπόν. Πρώτο και κύριο, πολιτική λύση στις συγκρούσεις. Εάν εξασφαλιστεί η πολιτική λύση, μπορεί να υπάρξει βελτίωση, ιδάλλως θα συνεχιστεί το πρόβλημα. Δεύτερο συμπέρασμα, πρότιμα ο άνθρωπος να έχει τη βοήθεια που χρειάζεται στη χώρα του ή σε μια γειτονική χώρα. Με αυτό λοιπόν διαπιστώνουμε ότι αν θέλουμε να πλησιάσουμε κάποιον και να του προσφέρουμε βοήθεια, Φερρυπίν, στη Γερμανία, αυτό θα κοστίσει 16 φορέ περισσότερο, οικονομικά σε οικονομικού όρου αυστηρά, από ότι αν του προσφέραμε την αντίστοιχη βοήθεια στον Λίβανο ή και στη Συρία ακόμη. Αυτό είναι άμεση συνέπεια τη ε, μετανάστευση. Επίση, περισσότερε από τι συγκρούσει αυτέ τραβούν όλο και περισσότερο στον χρόνο στον 7ο χρόνο τη είναι η σύγκρουση της Συρίας. Δηλαδή ένα παιδί που ήταν 6 ετών όταν άρχισε αυτή η σύγκρουση είναι τώρα έφηβος και γνωρίζει μόνο τη σύγκρουση. Έχει χάσει την παιδική του ηλικία, έχει χάσει κάθε ευκαιρία σε εκπαίδευση. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι Θυμάστε ότι σας είχα πει 9 στα 10, στις 10 χώρες ε, που πηγαίνουν μετανάστευση είναι χαμηλού και μεσαίου εισοδήματο. Ταυτόχρονα λοιπόν αυτοί που υποδέχονται τους μετανάστες οι χώρες, οι πολίτες, εξαντλούνται και οικονομικά. Όχι μόνο ο Λίβανος, η η Ορδανία, αλλά και η Ουγγάντα που δέχεται πρόσφυγες από τον Νότιο Σουδάν. Είναι οι κύριοι, κύριες χώρες προορισμού και υποδοχής ε, προσφύγων ή μεταναστών και εξαντλούνται όλο και προς το οι δυνατότητές τους. Και μια τελευταία σύσταση. γιατί διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι πρόσφυγες χρησιμοποιούν την ε, τεχνολογία, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να αναζητήσουν ε, προορισμό, τρόπο, δρόμο, δρομολόγιο ε, ή σύστημα που θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Όσο λοιπόν λιγότερο όσο λιγότερο ομοιόμορφα είναι αυτά τα, αυτές οι κινήσεις μετανάστευσης, τόσο διαφορετικές πρέπει να είναι και οι λύσεις που θα δοθούν. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο. Κάποιος που έφυγε πριν από τον υποψήφιο πρόσφυγα ε, θα τον ενημερώσει ποιο δρόμο να πάρει και πού να πάει. Σημαντικό για μας λοιπόν είναι να βρεθεί ένας νέος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί η ειρήνη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Τρεις αρχές, τρεις κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτον, μην φέρνει ζημία το σύστημα το οποίο θα σχεδιάζουμε. Μην κάνει κακό δηλαδή σε αυτούς που θέλουμε τελικά να βοηθήσουμε. Δεύτερον, οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα για την ε, εξασφάλιση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των ε, δομών, ταυτόχρονα πρέπει να προσφέρεται και η ανθρωπιστική βοήθεια για να διασωθούν ζωές ή περιουσίες. Και τρίτον, γιατί ξέρετε πολύ συχνά ε, αναφέρεται ότι οι τροφές, το τρόφιμα χρησιμοποιούνται και ως όπλα για τον πόλεμο, αποστερούνται δηλαδή τις τροφές οι άνθρωποι μέσα στι συνθήκε αυτέ. Ναι, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να γίνουν και όπλα για την ειρήνη, δηλαδή να προσφέρετε εγκαίρως η επιστηστική βοήθεια και να βοηθάτε και να βελτιώνετε ταυτόχρονα πολύ γρήγορα η κατάσταση. Τελευταία παρατήρηση. Είτε πρόκειται για Βόρεια, Ανατολική, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Σομαλία, η Πρώτα απ' όλα Πρέπει να γίνει λόγος για την ειρήνη, πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη. Μέχρι ότου όμως εγκαθιδρυθεί η ειρήνη, πρέπει πρώτον να εξασφαλιστεί ανθρωπιστική πρόσβαση σε αυτούς που υποφέρουν και μάλιστα βιώσιμη ανθρωπιστική ε, πρόσβαση και δεύτερον κατάλληλη χρηματοδότηση. Το ένα χωρίς το άλλο σημαίνει ότι είτε δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη με την ανθρωπιστική βοήθεια, είτε είναι υπερβολικά δαπανηρό σε βαθμό που δεν μπορεί να φέρει το απαιτούμενο αποτελέσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εξαιρετική ως και στο χρόνο σας. 10 λεπτά. Η Κριστίνα Μαράλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που ε, σας μιλώ εδώ σήμερα είναι η επίσημη ε, τελετή για την Παγκόσμια ε, ημέρα τροφίμων θα ε, γίνει στη Ρώμη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τα σπίτια τους και είναι πολύ πιο μεγάλος ο αριθμός τους από ότι οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτό ε, αναφέρθηκε οφείλεται σε συγκρούσεις και πολιτική αστάθεια βεβαίως. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει και ε, μια στρατηγική κατάλληλη για διαχείριση κινδύνων. Ε, η επισητιστική ασφάλεια, η ένδια, η έλλειψη ασφάλειας, έλλειψη θέσεων εργασίας, ανεργία ε, εξάντληση φυσικών πόρων, υποβάθμιση της γης ε, και ε, φυσικές καταστροφές όπως αυτές που είδαμε φέτος με την ξηρασία. Το 2015 είχαμε 244 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες, αλλά υπάρχουν και 763 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι μετακινούνται εντός των χωρών τους. Αυτές οι μεγάλες μετακινήσεις αποτελούν σύνθετες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν παγκόσμια δράση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έκανε τη διάσκεψη για τη διαχείριση της μετανάστευσης τον Ιούλιο του 2017 ε, επεσήμανε αυτή την ανάγκη να υπάρχει μια ε, συντονισμένη και παγκόσμια δράση. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στη συνέπεια της μετανάστευσης στις περιοχές της Υπέθρου ε, και στα νοικοκυριά της Υπέθρου και να πω ότι μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερα σε ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες. Γιατί τώρα τις περιοχές της Υπέθρου και γιατί τους νέους και τις γυναίκες. Τα τρία τέταρτα των εξαιρετικά φτωχών βασίζουν την βιωσιμότητά τους στη γεωργία και στις αγροτικές δραστηριότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν γη, που έχουν ένα μικρό κομμάτι γης, δεν μπορούν ε, να επιβιώσουν ε, και με τόσο μικρέ ε, όσα παράγει η γη τους. Και πολύ μεγάλο μερίδιο των μεταναστών προκύπτει από αυτές τις περιοχές της υπαίθρου. Έχουμε πάνω από 141 ε, ε, δις ε, δολάρια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα δίνονται για επιστημιστική βοήθεια και τελικά αυτά επιστρέφουν αλλού και όχι στους ίδιους τους μετανάστες. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι νέοι άνθρωποι και φυσικά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και κυρίως ανδρική μετανάστευση και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Γεωργία είναι γυναική υπόθεση. Ε, έγινε μια μελέτη πέρσι η οποία εξέτασε ε, τη δομή ε, των οικοκυριών και τις αγροτικές εργασίες και την ενδυνάμωση των γυναικών στη Γεωργία και κατέστη σαφές ότι σε πολλούς από αυτούς τους τομείς η υπεθρός γυράσκει και έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών και φτωχότερων ανθρώπων. Και επίση διαπίστωσα, ε, η σώμασε το ίδιο πράγματα όταν ταξίδεψα στον Νίγηρα και στο Μάλι. Υπάρχουν χωριά που είχε μόνο, είχαν όλο ηλικιωμένου γυναίκες και παιδιά. Και αναγκάζονταν φυσικά να δουλέψουν για τα προστοζήν, γιατί ορισμένες φορές οι άνθρες που ήταν μετανάστες δεν μπορούσαν να στείλουν χρήματα για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Η δομή λοιπόν και η αλλαγή ε, στις περιοχές της υπαίθρου είναι πάρα πολύ ε, σημαντική μοχλή μετανάστευσης. Επίσης, πρέπει να ε, επαγρυπνούμε, διότι αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αύξηση κατά 100 εκατομμύρια ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών που ε, θα αυξηθούν μεταξύ του 2015 και του 2030 και αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν ε, θέσεις εργασίας και ε, εισόδημα. Η μετανάστευση είναι ε, κοινή απάντηση ανθρώπων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ε, τις αντίξωες συνθήκες της ζωής τους. Ε, και επίσης είναι τμήμα της διαδικασίας της ανάπτυξης. Έχουμε δει ότι σε όλες τις οικονομίες που υπόκεινται διαθροτική ε, μετατροπή, η μετακίνηση ανθρώπων σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών ε, απασχόλησης είναι αναπόφευκτη και επομένως η μετανάστευση δεν θα εξαφανιστεί. Ε, επενδύσεις στον γεωργικό τομέα, στην αλυσίδα αξιών και στην ανάπτυξη της υπόθρου, πρόθεση της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης ε, θα βοηθήσουν Επίσης θα έχουμε και αύξηση στην ε, υποστήριξη της ανάπτυξης, τα δίκτυα μεταφορών, όλα αυτά δημιουργούν νέες ευκαιρίες για νέες δουλειές. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες για να υποστηρίξουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού όλα αυτά, αλλά και ε, τις κοινότητες που φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους, που πολλές φορές είναι και οι ίδιοι φτωχές ε, κοινότητες. Δεν υπάρχει ε, κάποια πανάκια βεβαίως, ε, δεν θα λύσει η ανάπτυξη τα πάντα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διασταυρούμενη προσέγγιση μεταξύ διαφόρων πολιτικών και φυσικά μια προσέγγιση για νόμιμη μετανάστευση η οποία φυσικά θα είναι και προς όφελος των χωρών προορισμού. Επιπλέον θα πρέπει να εξετάσουμε και την αλλαγή στις περιοχές της Υπέθρου, ιδιαίτερα στην Υποσαχάρη Αφρική, ως ένας βασικός παράγων ε, που καταδεικνύει ότι χρειάζεται κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι ε, θα πρέπει να επενδύσουμε σε αμυγός γεωργικές δραστηριότητες, αλλά ε, θα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλες δραστηριότητες. Μόνο όταν αλλάξει ο ιστός της υπαίθρου θα αλλάξουν τα πράγματα και οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή σε μικρές πόλεις, ε, μικρότερες των 500.000 ε, ε, ανθρώπων, μικρές κομοπόλεις και είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν τις αγορές των αργωτικών προϊόντων και συνδέουν τις αγορές με μεγαλύτερες αστικές περιοχές και εκεί μπορούμε να έχουμε και το επίπεδο συγκέντρωσης που οδηγεί σε παραγωγική γεωργία. Να επενδύσουμε λοιπόν στις κατασκευές και σε σύγχρονους τομείς. Σε πολλές χώρες ε, ε, όλα αυτά υστερούν και επομένως οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις περιοχές της υπαίθρου, προσπαθούν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον και τελικά απλώς διευρύνεται ο αριθμός ε, των φτωχών του άστεως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και φυσικά εάν δεν έχει γίνει τίποτα για να αλλάξουν αυτές οι τάσεις και αν δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, και δεν αλλάξει τρόπος ε, της γεωργίας στις παγκόσμιες αγορές, ε, την επόμενη δεκαετία μπορεί να έχουμε επιπλέον 1,7 δισεκατομμύρια άτομα τα οποία θα εγκαταλείψουν την γεωργία. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία και αυτά τα γεγονότα ε, είναι αυταπόδεικτα, μιλούν από μόνα τους, χωρίς να υπάρξει πραγματική αλλαγή στην προσέγγιση, στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Και μάλιστα ένας από τους ε, στόχους ε, της φετινής έκθεσης ε, για την γεωργία είναι να αναζητήσουμε και θεμελιώδεις στόχους. Τι εννοώ. Οι περιοχές της Υπέθρου είναι κάποιες περιοχές, αλλά δείχνουν και λίγο τον πολιτισμό. Πώς επιλέγουν τις τροφές τους, τι να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Έχουν και ένα αμυγός πολιτιστικό στοιχείο. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε περισσότερους δεσμούς μεταξύ των περιοχών της Υπέθρου και των μικρών πόλεων και κομοπόλεων που αποτελούν αυτή τη συνέχεια μεταξύ ε, του ιστού της υπαίθρου και της, ε, των αστικών περιοχών είναι αυτό το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες, ε, στον γεωργικό τομέα αλλά και σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες, σε μεταποίηση στον τομέα των μεταφορών, ε, θέσει εργασίας οι οποίες θα μπορέσουν να αποτελέσει λύση για να επιλέξουν κάποιοι να παραμείνουν στις χώρες τους. Του χρόνου η ΦΑΟ μαζί με το ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης θα προεδρεύσει στο Global Nation Group και θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την επιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη γεωργία στις κλιματικές αλλαγές και πώς μπορούμε να έχουμε συνθήκες μέσω των οποίων οι άνθρωποι να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα τους. Και επίσης ε, θα συνεχίσουμε με τους συναδέλφους ε, στο OMP ε, να δούμε τι σχέσεις υπάρχουν και με τις συγκρούσεις να πω ότι η μετανάστευση είναι τμήμα της διαδικασίας της ανάπτυξης και όπως οι οικονομίες υπόκεινται διαρθρωτικές αλλαγές, ο κόσμος θα μετακινείται. Η πρόκληση είναι να αντιμετωπίσουμε και τις οικονομικές πτυχές αλλά και τις κοινωνικές πτυχές, διότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ πολιτικών κοινωνικής προστασίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πιο φτωχούς ε, για να αναλάβουν κινδύνους και να ξεκινήσουν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα τους απομακρύνουν μεν από τα αγροκτήματα αλλά θα τους επιτρέψουν να έχουν μια καλύτερη ζωή στις περιοχές της υπαίθρου και σε αυτό το ε, συνεχές συνδετικό κρίκο που υπάρχει μεταξύ περιοχών της υπαίθρου και μικρών πόλεων. Και πρέπει να γίνει μία σύνδεση με τις περιοχές της υπαίθρου και αυτό φυσικά ε, θα είναι ιδιαίτερα υποφελές. Δεύτερον, η έγκριση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Επενδύσεων είναι βασικός παράγων, τον οποίο φυσικά επικροτούμε, διότι ε, θα υπάρχει και ανάγκη να γίνεται καλύτερη χρήση και των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών κονδυλίων με συνέργειες και με τρόπο ο οποίος θα συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, ε, στην εκρίζωση του θυμού και ε, της πείνας και φυσικά των βιώσιμων στόχων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, σας ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Θα ακολουθήσω το καλό σας παράδειγμα και δεν θα σας πλήξω μέχρι θανάτου με το PowerPoint. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω τις ήδη πλήρεις ιστορίες σας θα ήθελα λοιπόν να σας πω τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές από πλευράς Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαχείρισης Πολιτικών που είναι ο κόμβος μας και η απαρχή του εγγράφου που αφορά το πρόγραμμα μετανάστευσης και το πρόγραμμα διατροφικής ασφάλειας υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο. Άρα υπάρχουν τέσσερα βασικά ε, μηνύματα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργήσουμε υψηλές προσδοκίες όταν λέμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της ε, κακοδαιμονίας, της μετανάστευσης. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευφύς ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μακροχρόνιες και διαρθρωτικές επιπτώσεις της ε, διατροφικής ασφάλειας. Θα πρέπει να καλύψουμε επίσης το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και επίλυσης ε, διαφορών και θα πρέπει επίσης να προβάλλουμε συνολικές πολιτικές στο εμπόριο, ε, την αλληλεία, τα προγράμματα κατανάλωσης καθώς και την φορολόγηση. Η Κριστίνα είπε πολύ σωστά ότι η μετανάστευση είναι αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης καθεαυτής. Αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή. Το 2013 υπήρχε σοβαρή δέσμευση για τον ορισμό της πολιτικής μετανάστευσης ε, και η παγωγή της στην ανάπτυξη. Άρα βλέπουμε την μετανάστευση μέσα από αυτό το φακό της ανάπτυξης και αυτό ακριβώς έκαναν και οι συναδελφοί μου, αυτή την ανάλυση δηλαδή έκαναν ως προς τις επιπτώσεις στις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές χρηματοδότησης. Αυτή είναι μια πολύ καλή μελέτη, αλλά φυσικά θα πρέπει να δούμε και αυτό το σύνδεσμο της μετανάστευσης με την ανάπτυξη. Δεν έχω την ίδια πείρα με τους συναδέλφους και θα προσπαθήσω να εστιάσω σε ορισμένα ε, σημεία την παρουσίασή μου. Είναι πολλοί οι παράγοντες που οθούν στη μετανάστευση. Και όταν λέμε για, τις, ε, για τη ρίζα, για τα αίτια της μετανάστευσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία μας δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε περισσότερη μετανάστευση πριν βρεθούμε στο κάτω μέρος της καμπύλης. Τι λοιπόν έχει γίνει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Καταπίστευμα για στην Αφρική που ε, συστάθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτα το καλοκαίρι του 2015. για να χρηματοδοτηθούν 117 προγράμματα για 1,9 ε, δις ε, κατά 1,9 δις. και αυτό αφορά και την περιοχή του Σαχέλ. Μιλάμε για οικονομικά προγράμματα, ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών και της ασφάλειας και τις ε, κοινωνικές πολιτικές που μιλήσατε, την ε, υγεία, την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να έχουμε βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση στις χώρες προέλευσης. Ξέρουμε ποιες, είναι οι επιπτώσεις αυτών των προγραμμάτων εν μέρη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για τις διαρθρωτικές επιπτώσεις. Ε, έχουμε μελέτες του ECDPM και υπάρχει αυτή η δυναμική πορεία θετικών επιπτώσεων από την ενισχυμένη χρηματοδότηση για τομείς που βρίσκονται έξω από το στόχαστρο των ε, κυβερνήσεων και των φορέων χρηματοδότηση. Δηλαδή μιλάμε για όμορες περιοχές οι οποίες είναι εγκαταλειμμένες σχεδόν. Και εδώ βλέπουμε ότι Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ε, γίνεται σημαντική χρηματοδότηση για αυτόν τον τομέα στο κέρας της Αφρικής ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης. Θα δούμε όμως πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στους ευάλωτους αυτούς τομείς. Ιδιαίτερα στο κέρας της Αφρικής και, στην, ε, και στη, στη Σαχέλ. Γιατί εδώ έχουμε παραδοσιακά σχήματα μετανάστευσης που έχουν ε, μεγαλύτερη σημασία για την επιβίωση των μεταναστών. Μιλάμε λοιπόν για τα ολοένα και ε, διονγκούμενα αλλά και εναλλακτικά σχήματα μετανάστευσης και θα πρέπει να δούμε πόσο μπορεί να υπάρχει αρνητική επίπτωση στα παραδοσιακά σχήματα κινητικότητας. Βεβαίως ε, και αυτές οι πολιτικές ανοιχτών συνόρων θα μπορούσαν να σταθούν επιζήμιες πολλές φορές. Θα ήθελα να τονίσω και άλλα δύο σημεία. Υπάρχει αυτό το χάσμα γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και χρηματοδότησης εμείς ως δωρητές θα πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των οργανώσεων από τις χώρες εταίρους, αλλά και την ίδια την πολιτική των εταίρων μας, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα σε αυτά τα εγχώρια προγράμματα διατροφής. Γιατί υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια η οποία λειτουργεί πραγματικά από πάνω προς τα κάτω και απ' την άλλη ο ΦΑΟ που συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών φορέων. Θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντας τα εξής θα πρέπει να είσαστε πολιτικά ευφυείς υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή να μπορέσετε να επενδύσετε σε εγχώριους φορείς που έχουν ε, τη δυνατότητα να προβάλλουν αυτή την εδαφική προσέγγιση και επενδύσεις για καλύτερα στοιχεία από τις περιφέρειες. Επίσης, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο εύρος από τις επίσημες επισητιστικές πολιτικές που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίπτωση στη ε, ζωή και στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ όλους. Εξαιρετικές οι παρουσιάσεις σας. Και τώρα μπορούν οι βουλευτές να πάρουν το λόγο. Ελπίζω σύντομα οι ερωτήσεις. Μέχρι δύο λεπτά. Η κυρία Χόιμπλε. Ευχαριστώ πολύ. για τις ομιλίες σας. Ιδιαίτερα η τελευταία. Ψύχρεμη αντικειμενική μας έδειξε μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Και το ερώτημα πώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο ανθεκτικούς τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είπατε εσείς ότι στην Ήπεθρο και ιδιαίτερα οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο. Η γεωργία ασφαλώς ε, μπορεί να βοηθήσει. Στην πράξη όμως τι κάνουμε. Έχουμε την τάση να εξάγουμε το βιομηχανικό γεωργικό μας μοντέλο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό να είναι αίσθηση εργασίας. Αντίθετα, στην Ευρώπη έχουμε χάσει με την εκβιομηχάνηση της γεωργικής παραγωγής πολλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν όμως δυνατότητες για ε, λιγότερο εντατικές και ε, ολιστικές μεθόδους παραγωγής που δεν είναι οι βιολογικές ε, που θα μπορέσουν να δώσουν ένα διαφορετικό τόνο και λύσεις. Νομίζω ότι μέσα από τα προγράμματα αυτά πρέπει να προσφέρουμε τη γνώση και με ανταλλαγή τεχνονοσίας και με την έρευνα βεβαίως που θα πρέπει να διατεθεί για τους ανθρώπους αυτούς. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η συνοχή στην πολιτική που θα ακολουθούμε. Αναφέρθηκε και νωρίτερα. Δεν θα επιτύχουμε τίποτε εάν εδώ, στις χώρες αυτές, εάν εμείς εδώ κάνουμε το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε με άλλες πολιτικές μας. Όταν προσπαθούμε από την Ευρώπη να επιβάλλουμε στρατηγικές παγκόσμιας αγοράς και ενίσχυση των εξαγωγών, δεν μπορούμε να βοηθούμε τους ε, ανθρώπους στις χώρες αυτές. Ε, το, τα βιοκαύσιμα, παραδείγματι, μπορούν να αποτελέσουν ένα παράγοντα ο οποίος θα ανατρέψει τις πολιτικές για υποστήριξη της επιστηστικής ανάγκης. Ευχαριστώ, Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ σε μία πτυχή μόνο θα σταθώ. Κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές συγκρούσεων από την αρχή του χρόνου ξέρουμε ότι λείπουν 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια για τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες και κυρίως στο Νότιο Σουδάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Ξαναδιαβάζοντας ε, τα συμπεράσματα του G7 της Ταουρμίνα, το πρόβλημα είναι γνωστό, καταγράφεται και στα συμπεράσματα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έγιναν στην Ταουρμίνα, όπου ο Ιταλός Πρωθυπουργό μίλησε για την κρίση αυτή ε, αναφερόμενο στα 6 δισεκατομμύρια που χρειάζονται. Ο Τραμπ έβγαλε, πρόεδρος των ΗΠΑ, ε, έβγαλε τα ακουστικά του, δείχνοντας προφανώς ότι δεν θέλει να γίνεται λόγος, δεν θέλει πια να ακούει να γίνεται λόγος γι' αυτό. Ερωτώ λοιπόν, τώρα πού βρισκόμαστε, ποιο είναι ε, το επίπεδο χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Γιατί αν μαθαίνουμε ότι ε, λόγω της απουσίας της ε, έγκαιρης χρηματοδότησης κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, ερωτώ τους ειδικού μας τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτό το πρόβλημα και την ε, έλλειψη χρηματοδότησης για το μέλλον. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να βρεθεί μια μορφή χρηματοδο... προχρηματοδότησης για την ακρίβεια από ορισμένους φορείς όπως Φερρυπίν Παγκόσμια Τράπεζα που στη συνέχεια θα επέστρεφε τα ποσά αυτά ζητώντας την αναχρηματοδότησή τους από τα μέλη της. Μήπως θα μπορούσαμε έτσι να αποφύγουμε αυτήν την αποτρόπαια κατάσταση που πεθαίνουν της πείνας οι άνθρωποι επειδή δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές θα ακούσουμε την Επιτροπή, την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με τη σειρά, από ένα-δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Η Επιτροπή πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ από τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Θέλω να πω ότι είμαστε προσιλωμένοι στην, ε, και συμμετέχουμε στη συζήτηση αυτή για την επιστημιστική ασφάλεια, τις συγκρούσεις και τη μετανάστευση. Όχι μόνο όμως, δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο στη συζήτηση, αλλά δίνουμε και ταχεία απάντηση σε επιστηστικές κρίσεις που σημαίνει και πρόληψη και αντίδραση και ανα, ε, ανάκαμψη και ανικοδόμηση. Ε, από τα μέσα που διαθέτουμε θα σας αναφέρω δύο μόνο. Και βέβαια έχουμε ε, συνεργασία με WFP, την FAO και την ECO και θα αναφερθώ στην Παγκόσμια έκθεση για την επιστηστική κρίση, ετήσια έκθεση. Το 2018 θα εκδοθεί η τρίτη σχετική έκθεση και δίνει την, ε, ε, από το αποτύπωμα των επιστηστικών κρίσεων σε όλο τον πλανήτη. Μια κοινή μεθοδολογία χρησιμοποιείται, όπως και εταιρική σχέση με συνεργασία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της WFAO. Και επίσης πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφέρω ότι το 2017 η έκθεση καταγράφει 48 επιστηστικές κρίσεις, 11 χώρες πληττόμενες από συγκρούσεις και υψηλή αβεβαιότητα επιστηστική, οι τέσσερις κύριες επιστηστικές κρίσεις Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, η χώρες συγκρούσεως. Και το επόμενο εργαλείο που συνδυάζεται στην έκθεση αυτή με μια παγκόσμια αξιολόγηση των κρίσεων που ξεκίνησε από τους επιτρόπους στη Λιανίδη και Μίμητσα, WFP, FAO στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης. Το, το φόρουμ αυτό λοιπόν μπορεί να στηριχθεί στις πληροφορίες που δίνει το Global Report για να, η παγκόσμια έκθεση δηλαδή, για να ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η συζήτηση, αλλά και να εξασφαλιστεί ο συντολισμό και η διασύνδεση των μέσων που είναι απαραίτητη όταν μιλούμε για συγκρούσεις και επιστηστική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή υπάρχει και μια άλλη ομιλήτρια. Χαίρετε. Από την ΕΚΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά θα σας ήταν χρήσιμα κάποια νούμερα για την επιστηστική και διατροφική βοήθεια. Έχουμε ιστορικά το 50% του προϋπολογισμού της ΕΚΟ που πάει στην επιστηστική βοήθεια και διατροφική βοήθεια και για το 2016 917 συνολικά εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν στην ανθρωπιστική, επιστηστική και στη διατροφική βοήθεια που περιλαμβάνει και τις κτηνοτροφές ως βοήθεια με κύριο εταίρο μας την WFP αλλά και την FAO μεταξύ των 11 εταίρων μας για την επιστηστική βοήθεια και για να δώσω απάντηση στην ερώτηση τη σχετική με τις χώρες ε, που κινδυνεύουν από λοιμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δική μας Γενική Διεύθυνση μαζί με τους συναδέλφους της ΔΕΦΚΟ ξεκίνησαν από την αρχή του χρόνου την κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τις χώρες αυτές, για την Ιγυρία, παραδείγματι, και την περιοχή της λίμνης Τσάντ, συνολικά 105 εκατομμύρια για την αναπτυξιακή και πιστιστική βοήθεια, η Σομαλία 120 εκατομμύρια, το Νότιο Σουδάν και η γειτονική περιοχή 250 εκατομμύρια, η ΔΕΗ εμένη 116 εκατομμύρια. Είναι τα ποσά τα οποία χορηγήσαμε για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια εν ολίγης. Επίσης, η προσέγγιση, η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι μια ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο και την ανοικοδόμηση των τοπικών κοινωνιών. Στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε συστήματα ενημέρωση για την ασφάλεια των τροφίμων και προειδοποίησης και βέβαια οι συνάδελφοι από την ΕΦΕΟ μας βοηθούν ιδιαίτερως. Η δε ανθρωπιστική βοήθεια, όπως γνωρίζετε, είναι πάντα ανεξάρτητη, ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές και προσφέρεται αναλόγως των αναγκών. Είναι όμως περιορισμένες οι δυνατότητές της. Κυρίως σε περιοχές συγκρούσεων Γιατί όσο δεν υπάρχει πολιτική λύση στην κρίση, όσο και να προσφέρουμε εμεί τη βοήθεια, μόνο θα χρειάζεται παραπάνω βοήθεια, λύση δεν θα δίνεται. Και για δύο λεπτά μόνο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τη δική μας την ε, θέση και συμμετοχή. Ε, υπενθυμίζω ότι το τελευταίο μόνο μήνα κάναμε πάρα πολλά. Επί παραδείγματι, συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον εξορθολογισμό της διασύνδεσης αναπτυξιακής βοήθειας και κοινή ανακοίνωση, κοινό ανακοινωθέν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στρατηγική προσέγγιση για την ανθεκτικότητα και στη χρήση της εξωτερικής δράσης, 7η Ιουνίου. Ιδιαίτερα το κοινό ανακοινωθέν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εξετάζει ε, με ευρύτερο πρίσμα την ε, ενίσχυση της ανθεκτικότητας Και έτσι καλύπτει όχι μόνο την ασφάλεια ή απουσία ασφάλειας τροφίμων, αλλά και την κοινωνική διάσταση, το πώς είναι οι κοινωνίες αυτές. Και έτσι έχουμε απαντήσει και για το πώς μπορούμε να αντιδρούμε ή τι είδους στρατηγικές πρέπει να αναπτύσσουμε για το μέλλον. Χρειάζεται βέβαια μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, μια πιο ολιστική προσέγγιση μεταξύ της ανθρωπιστικής και της ε, αναπτυξιακής ε, βοήθειας, αλλά βέβαια και η δυνατότητα να συναντηθούν όλοι οι παράγοντες στο τραπέζι των συστήσεων. Στο Ταλίν, στο άτυπο συμβούλιο, υπήρχε η ευκαιρία για συζήτηση. Ε, χώρες ανέλαβαν πιλωτικά τη δοκιμή, τη δοκιμασία, ε, τη δοκιμή μιας νέας ε, προσέγγισης για τη διασύνδεση και πρόκειται για το Σουδάν, την Ουγκάντα, την Νιγηρία, την Μιανμάρ, το Ιράκ και άλλη μια χώρα, έκτη χώρα την οποία δεν βρίσκω και το Τσάντ Εξετάζουν λοιπόν τη διασύνδεση μεταξύ ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. και τώρα συζητούμε με τις αντιπροσωπείε μας τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην κάθε περιοχή. Θα είναι βέβαια προσέγγιση μέσω των κυβερνήσεων, αλλά πάνω από όλα μας ενδιαφέρει να επιληθούν ή να δοθεί βοήθεια στην επίλυση αυτών των κρίσεων ε, με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ευχαριστώ και τώρα θα απαντήσει το πάνελ με αντίστροφη σειρά. Πρώτα η κυρία Μολίνα. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για όλα σας τα σχόλια στις παρουσιάσεις μας και θα ήθελα να επισημάνω και κάποια θέματα τα οποία συζητήθηκαν, τι άκουσα. Ο πρώτος ομιλητής ε, πολύ σωστά επεσήμανε την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των κρατών μελών ε, της Ένωσης να επενδύσουν ε, σε διαρθρωτικές λύσεις για την ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών συστημάτων διατροφής, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα μακροπρόθεσμου οράματος, το οποίο πρέπει να επιδείξει και μια πολιτική ευφυΐα. Να δούμε ε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και τους τοπικούς παράγοντες στις δυνατότητες παρέμβασής τους. Δηλαδή να μην έχουμε κατά νου μόνο ε, διεθνείς ερευνητικούς φορείς, αλλά να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε σε τοπικό επίπεδο και τους μικρούς γεωργούς με τις αρμόδιες υπηρεσίες που ορισμένε φορές είναι αποδυναμωμένες και με εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά εκεί ε, έχουμε και την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και ε, το πρόβλημα στη ρίζα του για την επιστημιστική ασφάλεια. Ε, με τα χαρά άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ε, συγκεντρώσει γύρω από ένα τραπέζι όλους τους αρμόδιους φορείς ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και, και ε, ε, αναπτυξιακής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να τα πω από το πρίσμα της βιωσιμότητας. Ε, ποιο είναι το μοντέλο ε, γεωργικής ανάπτυξης που θέλουμε στο μέλλον. Το 85% των εκμεταλλεύσεων ε, ανά τον κόσμο έχουν λιγότερους από δύο ανθρώπους. Και αυτό κυρίως στην Υποσαχάρη Αφρική και στην Ασία. Εκεί έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα, αλλά έχουμε μεγάλη παραγωγικότητα της γης, που σημαίνει ότι τα μοντέλα του παρελθόντος, τα οποία είχαν ε, μεγάλη ένταση σε ενέργεια, σε νερό, δεν μπορούν να συνεχιστούν σε ένα σύστημα που ο κόσμος ε, ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, φτάνει και στο πέρας κάποιων ε, παραγωγικών δυνατοτήτων. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα θέματα πρόσβασης της γης. Σήμερα ο Επίτροπος Μίμητσα με το Γενικό Διευθυντή στη Ρώμη γιορτήσαν την πέμπτη επέτειο για την εθελοντική πράξη για τη γη. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Είναι μια ισότιμη διαδικασία που είναι, πρέπει να είναι προς όφελος όλων, όχι μόνο μερικών. Γιατί αν δεν υπάρχει ισότητα με μεγαλύτερη παραγωγικότητα στη γεωργία και καλύτερη χρήση της γης, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Πάντα θα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα περιθωριοποιούνται, που θα είναι φτωχοί ε, των αστικών περιοχών και θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γη τους. Ε, τα συστήματα λοιπόν ε, γεωργίας έχουν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις ε, τη σήμερα ημέρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε γνώσεις, να επενδύσουμε σε πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές και εδώ οι οργανώσεις των παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο διότι βεβαίως σε αυτό τον ιστό ε, άστεως και περιοχής της Υπέθρου θα πρέπει να αναζητήσουμε και νέους τρόπους ε, να ε, φτάσουν πιο κοντά οι καταναλωτές στους παραγωγούς. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε και τη γεωργία ως πολιτισμό από τη γη στο πιάτο σας και φυσικά τη διατροφική αξία της γεωργίας η οποία ε, θα έχει και σημαντικά ωφέλη γιατί θα προσφέρει καλύτερη υγεία του πληθυσμού και βεβαίως να ε, εξετάσουμε και το θέμα της ε, αποταμίευσης, ε, να μην σπαταλούμε νερό, να μην σπαταλούμε ενέργεια και να χρησιμοποιούμε και διαφορετικές τεχνικές. Όλα αυτά απαιτούν γνώσεις, απαιτούν εκπαίδευση, απαιτούν και διαφορετικές δεξιότητες και σήμερα πιστεύουμε ότι η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να φέρει όλες αυτές οι γνώσεις πολύ πιο κοντά στους γεωργούς από ό,τι στο παρελθόν. Εξετάζουμε λοιπόν αυτά. Και τέλος ο κύριος Χουσέιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Ε, είμαι οικονομολόγος και γι' αυτό θα σας δώσω αριθμητικά στοιχεία. 27 δις ευρώ το 16 για ανθρωπιστική βοήθεια 40% λιγότερα από τις πραγματικές ανάγκες. Από τα 27 δις δολάρια το 15% πήγε σε πέντε χώρες, Συρία, Ιράκ, Ιεμένη, ε, Αιθιοπία και μια άλλη χώρα και στο, το επόμενο 50% πήγε σε τρεις χώρες. για να καλύψει ανάγκες από 5 έως 95% στις χώρες αυτές. Ήταν η τέταρτη συνεχής αύξηση κονδυλίων, άρα χρήματα εισραίουν, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με περιοχές σειράξεων. Ως προς το δεύτερο σας ερώτημα, όταν δούμε τους αριθμούς ως προς την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπήρξε μεγάλη αύξηση πόρων μεταξύ 15 και 16, 2015-16. Ε, δηλαδή μιλάμε για 800 ε, εκατομμύρια δολάρια. Και από πλευράς ΕΠΑ έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα φέτος από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ δίνουν χρήματα όμως, όταν έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες, ε, φυσικά ε, φαινόμενα, η ξηρασία, αντί για όλα αυτά έχουμε να κάνουμε με περιοχές σειράξεων και αυτό δεν ξέρουμε πότε θα λήξει. Άρα νομίζω ότι η πορεία μας δεν είναι σωστή ως προς το στόχος βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030 αν δεν επιληθούν αυτές οι σειράξεις. Μιλάμε για 13 χρόνια μετά. Και γι' αυτό ο απαράβατος όρος είναι επίλυση διαφορών και σειράξεων. Και στη συνέχεια η επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ ε, λυπάμαι που σας έδωσα τόσο λίγο χρόνο. Οι παρουσιάσεις σας ήταν ε, εξαιρετικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα τελειώνουμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και τώρα φτάνουμε στο 16 ε, Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης στην Ονδούρα. Η επικεφαλής, η Λόλα Σάντσες, θα λάβει το λόγο και θα μας ε, δώσει, θα μας κάνει μια παρουσίαση και μπορούν και οι άλλοι αντιπρόσωποι να λάβουν το λόγο στη συνέχεια. Η Λόλα καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας κάνω μία συγκεφαλαίωση της αποστολής στην Ονδούρα. Η Ελένη Θεοχάρους ήταν μαζί μου καθώς και ο Ντόρου Φρουντσουλίκα. Η Ονδούρα είναι η πιο φτωχή χώρα της υπηρετικής Λατινικής Αμερικής και παρά το γεγονός ότι έχει 8 εκατομμύρια, ε, έχει χαμηλά εισοδήματα. Έχει πολλές, ε, πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσει για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα ως προς τις ε, ε, ως προς τις εξαγωγές και εισαγωγές και ιδιαίτερα ως προς την εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων και στον, ε, τον κλώστο υφαντουργικών. Υπάρχει ατιμορρησία, μεγάλη εγκληματικότητα και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο που έχει οδηγήσει και σε ε, θάνατο, θανάτωση ακτιβιστών τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων το 2016 δύο μεγάλων ακτιβιστών. Και μετά από τη Βολιβία έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες ε, μάστιγες σε τομείς όπως δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική ισότητα και αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών. Και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βελτιωθούν όλα αυτά. Είχαμε ένα εντατικό πρόγραμμα δύο ε, ημερών. Συναντηθήκαμε με την, ε, με την Αντιπροεδρία του Κογκρέσου και εκπροσώπους της κυβέρνησης, διεθνείς οργανώσεις συνεργασίας στην ανάπτυξη, διεθνείς οργανώσεις ΜΚΟ, καθώς και οργανώσεις γυναικών και ε, αυτοχθόνων, καθώς και διεθνείς ε, δωρητές και τον πρέσβη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της απαστολής είναι τα εξής. Υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί η ανθρωποκτονία, η εγκληματικότητα, η ατιμορρησία και ούτω καθεξής. Η έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η φοροδιαφυγή που υπάρχει σε πολλούς τομείς και πολλές φορές υπερβαίνει και το 70%. Η αναπτυξιακή συνεργασία έχει μεγάλη σημασία και τα μέλη της αντιπροσωπείας το τόνισαν αυτό. Δυστυχώς παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις υπάρχει διαφθορά και ατιμορρησία στη χώρα και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και συνεργασία, ιδιαίτερα ως προς τους ε, ευάλωτους γυναίκες, μετανάστες, ΛΟΑΔ δημοσιογράφους και ούτω καθεξής. Υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας καθώς και η πρόσληψη νέων ανηλίκων για τη διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά και πολλοί άλλοι τομείς διαφθοράς. Είναι απαράδεκτος ο είναι απαράδεκτες οι ε, δολοφονίες γυναικών. 40 γυναίκες ε, δολοφονούνται κάθε μήνα, το οποίο σημαίνει μία ε, δολοφονία κάθε στην ουσία 18 ώρες. Και ένα 12% ανηλίκων γυναικών έχουν υπάρξει έγκυες μετά από βιασμό ένα 12%. Και ως προς την βία στα πανεπιστήμια, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ε, δολοφονήθηκαν 42 ε, φοιτητές, 45 εργαζόμενοι και γύρω στους 50 εργαζομένους του δημόσιου τομέα και της ασφάλειας και έχουν σκοτωθεί συνολικά δολοφονηθεί 47.000. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα 70% δείκτης ατιμορρησίας σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια που προέρχεται από την αστυνομία γιατί χρησιμοποιούν βία και πολλές φορές υπάρχει και συμπεγνία με το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν πολλά πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα. Και δυστυχώς επιτρέπει η νομοθεσία να κατέχει ένας άνθρωπος πέντε όπλα. Επίσης η κατάσταση στο περιβάλλον είναι απαράδεκτη, καθώς και η κατάσταση των ΛΟΑΔ. Γίνονται δολοφονίες καθημερινά. Επίσης είδα μεγάλη βία από πλευράς ε, ΜΜΕ γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η εκπαίδευση και γι' αυτό δεν επιτρέπεται κάθε ώρα της ημέρας να βλέπει κανείς τα πτώματα και τις δολοφονίες όλες τις ώρες του 24ωρου και αυτό είναι απαράδεκτο για τα μικρά παιδιά, διότι τα μικρά παιδιά συνηθίζουν να βλέπουν αυτές τις εικόνες ε, σαν να επρόκειτο για ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε ένα 30% αλφαβητισμού και από όλες τις ε, πλευρές με τους συνομιλητές είχαμε ε, μία ευρεία συζήτηση ως προς την οικονομική και, κοινωνική κατάσταση, κάτι το οποίο φυσικά δημιουργεί σε σύγχυση. Βρισκόμαστε ενώπιον εκλογών. Έγινε λόγος για την νομιμοποίηση της άμβλωσης, η οποία ποινικοποιείται και για τις δημόσιες ελευθερίες. Χρειάζεται λοιπόν ένας πολιτικός διάλογος για να δημιουργούν συνέργειες και να αναπτυχθεί η χώρα. Η Ονδούρα δεν έχει εφαρμόσει καμία από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις εκλογές και πολλοί μίλησαν για ανησυχίες εάν επανεκλεγεί ο πρόεδρος μετά από την μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι δωρητές θα πρέπει να κρατήσουν αυτή την πίεση προς τη χώρα έτσι ώστε να γίνει μία αλλαγή ουσίας, έτσι ώστε να απομακρυνθούμε από τον ολοκληρωτισμό. Στο κοινωνικό επίπεδο, με βάση την, την εργασία της νέας ΟΚΕ, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου. Επίσης, Υπάρχουν πολλές ε, μεταρρυθμίσεις που δεν ε, είναι αποδοτικές επειδή δεν χρηματοδοτούνται. Αυτό αφορά και τους ανθρώπινους πόρους και τις ε, διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή υπάρχουν μεταρρυθμίσεις επί χάρτου, οι οποίες όμως δεν τίθενται σε εφαρμογή. Πολλά θα πρέπει να γίνουν, αλλά θεωρούμε ότι η δημοσιονομική υποστήριξη θα πρέπει να συνάδει και με τα προγράμματα τα συμπληρωματικά προγράμματα ή τα συνοδευτικά προγράμματα. Αυτό αφορά και την ε, επισητιστική ασφάλεια καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου φτάσαμε σε απτά αποτελέσματα. Υπάρχει ένας νόμος για να προστατεύει ΜΜΕ, δημοσιογράφους, ακτιβιστές και τη δικαιοσύνη που συντάχθηκε με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και δεν υπάρχουν και πόροι. Επίσης ε, υπάρχει στάση συνεργασίας με τις αρχές, ιδιαίτερα ως προς τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει μια συνεργασία υψηλού επίπεδου και ένα ε, γραφείο, καθώς και συνεργασία με την ΚΝΟΥΡ για να βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους, διότι υπάρχουν 170.000 εσωτερικά εκτοπισθέντες που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους. Ως προς την Συμφωνία Σύνδεσης ισχύει ο εμπορικός πυλώνας και θα πρέπει να υπάρξουν σωστές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη Συμφωνία 179 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Υπ' αυτή την έννοια γίνονται ε, συζητήσεις μέσα στα πλαίσια και της δικής μας ε, αποστολής για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αυτόχθονες. Τέλος, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Πασκάλ και Χουαν Κάρλος από τη Γραμματεία για την εξαιρετική τους εργασία και για την προετοιμασία αυτής της αποστολής. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε Λόλα. Η Ελένη Θεοχάρους έχει το λόγο. Couple Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτα πρέπει να συγχαρώ την ε, Λόλα όχι μόνο για την εξαιρετική ε, έκθεση που έχει καταθέσει αλλά και για τον τρόπο που διεύθυνε την αποστολή. Η Ονδούρα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα με εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση, επικίνδυνη αλλά με ένα πολύ έξυπνο λαό τουλάχιστον στον βαθμό που ε, μπόρεσα να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους. Είναι ένα λαός με ένα υψηλό IQ. Τώρα, οι παρατηρήσεις μου δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα στην ε, έκθεση, μάλλον δεν θα προσέθετα τίποτα. Κάποιες πιο γενικέ και κάποιες πιο ειδικές παρατηρήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ε, ή να σας είναι χρήσιμες. Η διαφθορά και η ατιμορρησία είναι το κυρίαρχο στοιχείο και με αυτή την έννοια επιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δίνει τεράστια κονδύλια όπως αυτά που δίνονται στην Ονδούρα είναι η δεύτερη ο δεύτερος ε, αποδέκτης κονδυλίων στην ε, Λατινική Αμερική μετά την Βολιβία, θα πρέπει να ασκεί και μεγαλύτερο έλεγχο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι σίγουρη αν όλα τα κονδύλια διατίθενται για τον σωστό τρόπο. Επίσης, ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα της διάθεσης της βοήθειας προς την κοινότητα κατευθείαν είναι κάτι για το οποίο επιμένω για χρόνια και όχι μέσω κάποιας διεφθαρμένης αρχής κυβέρνησης ή τοπικής κυβέρνησης, είναι αυτό που ζήσαμε σε μια δασική βιομηχανία όπου η κοινότητα ολόκληρη είναι εμπλεκόμενη σε μια συνεργατική βάση για την παραγωγή ε, ξύλου και την εκμετάλλευσή του και όλων των παραπροϊόντων που μπορούν να προκύψουν καθώς επίσης και κάποιων, ας μου επιτραπεί όρος, παρασιτικών ε, εκδηλώσεων που μπορεί να να δοθούν. Είναι μια, ε, ένα εξαιρετικό παράδειγμα σωστής διαχείρισης, αλλά δεν ισχύει αυτό σε όλη την έκταση. Όσον αφορά την κλωστοϊφαντουργία, που είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδημάτων, ε, εκείνο που άκουσα και με έχει σοκάρει, ακόμη και αν είμαι ένας σκληροτράχυλος γιατρός, είναι ότι οι άνθρωποι ε, μπορεί να κάνουν την ίδια μέρα μέχρι και 60.000 φορές την ίδια κίνηση αυτοί που εργάζονται στην γλωστοϊφαντουργία. Με αποτέλεσμα, όταν μπαίνουν στην υπηρεσία από τα 18 χρόνια, στα 30 να μην μπορούν πια να δουλέψουν. Να είναι εντελώς ε, medical unfit. Ε, επίσης, εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πολλά μικρά παιδιά κατά παράβαση του διεθνούς νόμου εργάζονται στην κλωστοϊφαντουργία και αυτό δημιουργεί όλες τις ε, συνέπειες, ε, ε, τις αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή τους. Όταν ερωτήσαμε τον εκπρόσωπο των βιοτεχνών και των βιομηχάνων για τις επαγγελματικές ασθένειες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην κλωστοϊφαντουργία, γιατί ήδη γνωρίζαμε κάποια πράγματα, μας απάντησε ανοήτως ότι πάσχουν από γρήπη, από κρυολόγημα, από ε, οτίτιδες, ενώ Ευτυχώς δεν μας είπε ότι και οι γυναίκες they do menstruate, εν πάση περιπτώσει. Ε, όταν ερωτήσαμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων, μας είπαν ότι, ε, δεν, το, δεν το δώσανε με ιατρικούς όρους, αλλά μας είπαν ότι πάσχουν από φρακτική πνευμονοπάθεια, από μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και από α, άλλες νόσους φθοράς, κυρίως των πνευμόνων ίσως από την εισπνοή των ινών. Καταλαβαίνετε ότι όταν τολμούν οι άνθρωποι να κάνουν αυτές τις καταγγελίες, πόσο πιο χειρότερη είναι η κατάσταση. Η τελική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό που έχει τονίσει και η Λόλα, ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία, γιατί μόνο οι άνθρωποι που ξέρουν δεν μπορούν να γίνουν υποχείριο του οποιοδήποτε και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όπως σας έχω πει το παράδειγμα της ε, μικρής κοινότητας που επισκεφτήκαμε και δεν θυμάμαι το όνομα της αυτή τη στιγμή είναι ε, ε, εξαιρετικό. Επίσης, εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα περίθαλψης και υγείας, είναι σκόρπια εδώ και εκεί κάποιος γιατρός ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εάν στηριχτούν οι επιστήμονες της χώρας να παραμείνουν και να να υπηρετούν στη χώρα τους τουλάχιστον πέντε χρόνια, εφόσον πολλοί σπουδάζουν με υποτροφίες, το αντάλλαγμα, το ανταποδοτικό που θα δώσουν σε αυτό που τους προσφέρει την υπηρεσία είναι να μείνουν πέντε χρόνια στον τόπο τους να δουλέψουν. Αυτό ήταν μια πρακτική που εφάρμοζε η Βρετανική Κοινοπολιτεία και από το οποίο εποφελήθηκα και εγώ. Γιατί, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, εμείς γεννηθήκαμε Βρετανοί. Δεν ξέρω αν θα πεθάνουμε Έλληνες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Σάχλ, θέλεις το λόγο. Ναι, είχα τη χαρά να ενημερωθώ από τη Λόλα και τη συνάδελφο που μίλησε μόλις τώρα για την επίσκεψή τους. Είναι, πιστεύω, σημαντικό το ότι έγινε αυτή η επίσκεψη και ότι μπορέσετε να συλλέξετε τόσες γνώσεις και πληροφορίες. Ο πρόεδρος, δύο, τρία συναδελφοί στον το λόγο, η υπηρεσία εξωτερική δράση, η ΔΕΦΚΟ και ο πρεσβευτής. Η υπηρεσία εξωτερική δράσης δεν θα μακρηγορήσω πρόεδρε. Είναι πολύ χρήσιμη έκθεση. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι μπορέσαμε να συμβάλλουμε ε, αποτελεσματικά στην προετοιμασία της ε, αποστολής. Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω ένα μήνυμα το οποίο απορρέει από την έκθεση αυτή ότι είναι αλληλένδετος ο αγώνας για την καταπολέμηση της, ε, του λοιμού, της πείνας και αυτός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται άλλωστε και για τη ραχοκοκαλιά τη δική μα δράση, όχι μόνο στην Ονδούρα, αλλά σε κάθε τομέα δράση μα. Η προαγωγή και ο σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων αναφερθήκατε στον Κάρσερε και βέβαια παρακολουθούμε και εμεί τι εξελίξει και βέβαια τη δίκη. Ε, τι, όταν ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την αντιμετώπιση της, ε, της των δασών, όλα αυτά βοηθούν την κοινωνία και πιστεύουμε ότι οι βουλευτές που ήταν στην αποστολή έγιναν μάρτυρες της προσπάθειας και της δράσεώς μας. Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της ε, FLECTVP, της συμφωνίας FLECTVP που αναφέρθηκε και νωρίτερα, ε, είναι μια συμφωνία όχι εμπορικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την πραγωγή της καλής διακυβέρνησης και δείχνει ότι μπόρεσε για πρώτη φορά να μπει σε ε, πρώτη προτεραιότητα το θέμα της ε, χρηστής διακυβέρνησης ε, και βέβαια όπως ζητούν και από την οργάνωση, παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας και το άρθρο 69 η ενημερωμένη συνένεση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει αρκετή πρόοδο, σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό της Ονδούρας. Ευχαριστώ. Εντεύχω τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εμεί θέλουμε να καλωσορίσουμε την έκθεση, η οποία σημειώνει βεβαίως ότι η όλη κατάσταση έχει βελτιωθεί, ότι η αναπτυξιακή συνεργασία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το διαβάζουμε με ικανοποίηση στην έκθεσή σας. Βεβαίως παραμένουν οι προκλήσεις. Βεβαίως συμφωνούμε ότι δεν έχει έρθει η ώρα να πενταπαθούμε στις δάφνες μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις εξελίξεις του τομείς ε, ε, που επισημαίνουμε όχι μόνο στη συγκεκριμένη έκθεση για την αποστολή σας αλλά στην ετήσια έκθεσή μας για το κράτος δικαίου και όλους τους ε, εγκάρσιους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, καταστολή, καταστολής της διαφθοράς και το καθεξής από την κίνηση αυτού του πλαισίου συνεργασίας του 2014 έχουμε ιδιαίτερα σταθεί σε αυτούς τους τρεις τομείς, αλλά κοιτούμε και τους εγκάρσιους τομείς, όπως είπα, το πρόγραμμα EuroAct, παραδείγματι, που ξεκίνησε πρόσφατα να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη έμφαση, αποκλειστική έμφαση στην καταπολέμηση διαφθοράς. Και συμφωνούμε με την ε, τοποθέτηση που διαβάζουμε στην έκθεση για τη σημασία του διαλόγου για την πολιτική και τη μεταρρύθμιση του δημόσιου, του συνθήκων δημοσίου διαλόγου. βεβαίω θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και βέβαια και η χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό διάλογος για την πολιτική είναι κομμάτι αυτής της χρηματοδότησης, Παρακολουθείτε η υλοποίησή του για ενόψη της χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη πολιτικών επίσης, όπως παραδείγματι στον χώρο της απασχόλησης, είναι στοιχείο που εξετάζουμε. Ο πρόεδρος ζητούσε, συγγνώμη που σας πιέζω τόσο για με το χρόνο, ο κύριος Τσόα, πρεσβευτής της χώρας για δύο λεπτά μόνο και βεβαίως αν θέλετε πιο πολλές πληροφορίες γραπτώς μπορείτε να μας στείλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής. Ε, καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Επιτροπής σας και για την ε, ε, αποστολή στην οποία επικεφαλής ήταν η κυρία Λόλα Σάνσε στην Ονδούρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την έκθεση που ακούσαμε σήμερα, ιδιαίτερα τις πολιτικές αξιολογήσεις τις οποίες σεβόμαστε αλλά δεν συμμεριζόμαστε. Θεωρούμε όμως ότι είναι επικοδομητική και γόνιμη διαδικασία και επίσης ε, δείχνουν ε, την εξαιρετική σχέση σεβασμού, επικοινωνίας και ανοίγματο ε, σε σχέση με την Ονδούρα. Η Ονδούρα είναι μια χώρα ανοιχτή για όποιον θέλει να πάει εκεί, όπως είπε η κυρία Σάντσες. Επίσης, ε, γνωρίσατε τις ε, εθνικές μας αρχές ε, που αμέσως σας έδωσαν πρόσβαση και μέσω και της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων ξεκίνησε μια διαδικασία μελέτης και απάντησης όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση. Ε, να είστε βέβαιοι ε, από την Επιτροπή σας ότι η κυβέρνηση και η Δημοκρατία της Ονδούρας ε, θα λάβει υπόψη της όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Αλλά δεν μπορώ να σταθώ μόνο εδώ. Θα πρέπει να πω και κάτι για την επικοδομητική θετική στάση που βλέπω και ως πολίτης του κόσμου αλλά και ως πολίτης της Ονδούρας. Η κατάσταση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια και η αναγνώριση των προσπαθειών για την πολύ σημαντική ε, μείωση του ποσοστού των ανθρωποκτονιών που αναφέρθηκε και η μείωση ε, ξεκινάει και με την συνεργασία για την ανάπτυξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βελτιώθηκαν κάποια κοινωνικά θέματα χάρη στι θετικές εργασίες τη ΕΟΚΕ, η οποία συστήθηκε χάρη στην υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω αναφέρθηκε. Χαιρόμαστε για την αναγνώριση ε, μετά από διαπραγματεύσεις της Συμφωνία Σύνδεσης Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και την κύρωση αυτή τη σύμφωνη. Ε, με όλες τις κοινότητες για να βρούμε και μια εθνική συνένεση για την υπογραφή της συμφωνίας. Και επίσης υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία. Συμφωνούμε την παρατήρηση της έκθεσης ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί πολύ καλό συνδυασμό κοινωνικού διαλόγου, συνεργασίας για την ανάπτυξη, ε, διαχείριση των δασών κλπ. Και κάτι επιπλέον θετικό. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή ΔΕΒΕ δέχτηκε με ικανοποίηση τη συμφωνία ω πνεύμα συνεργασία μεταξύ των φορέων τη Ονδούρα και δείχνει ότι ο διάλογο μεταξύ των πολιτών τη Ονδούρα είναι προ όφελο όλων. Το ξέρω ότι έχω 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσω. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ονδούρα είναι κάθε φορά όλο ένα και πιο ικανοποιητική. Είναι το τελικό συμπέρασμα το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα. Δεν θα ήθελα μόνο να σταθώ σε αυτό. Υπάρχουν και οι προκλήσεις και οι προκλήσεις ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ε, ε, άμεση συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε βοήθεια σε διάφορες πτυχές που αναφέρθηκαν και στην εκλογική διαδικασία και σε άλλες. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες προκλήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχω επαρκή χρόνο για να το κάνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα τα στείλω γραπτό στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λόλα, σας ευχαριστώ για την επίσκεψη. Να ευχαριστήσουμε και τους άλλους βουλευτές για την ε, επίσκεψη. Ε, συμφωνώ ε, με κάποια και διαφωνώ βεβαίω και με κάποια, αλλά είμαστε εδώ για επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την πολύ αποτελεσματική σας παρέμβαση. Λόλα, θέλετε να επανέλθετε. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώθηκε. Και τώρα θα αναλάβει και πάλι την Προεδρία η Λίντα. Θα μείνω εδώ, δεν χρειάζεται να μετακινηθώ γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά, ε, γιατί στις 5 πρέπει να φύγουμε για να πάμε να ψηφίσουμε. Έχουμε δύο ακόμα εκκρεμότητες, ε, αλλά η Τζούντι Αρζεντίνη απουσιάζει. Ε, είδα την ερώτησή της, έχουμε δύο προφορικές ερωτήσεις, έχουμε χρόνο. Ε, και για την ε, επόμενη συνεδρίαση. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να τις προτείνουμε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά γιατί δεν είναι εδώ. Θα γίνει η ερώτησή της λοιπόν την επόμενη φορά. Η κυρία Χόιμπουχ λοιπόν έχετε την ερώτηση εδώ αφορά την Επιτροπή του ΣΑΝΤΑΚ. Ε, σε μια συνεδρίαση πριν από το καλοκαίρι συζητήσαμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καθορίσει τη διαπραγματευτική στη θέση για την Επιτροπή ΝΤΑΚ για την αναπτυξιακή βοήθεια. Παρακαλώ λίγο ησυχία. συνεδριάζει στις 30 και 31 Οκτωβρίου η Επιτροπή ΔΑΚ, η συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τη θέση της για τη συνεδρίαση αυτή. Παρακαλώ, δεν έχω και το όνομα του εκπροσώπου. Νικολέτα Μέρλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πει την ημερήσια διάταξη τη 51 η συνεδρία τη υψηλού επίπεδου τη Επιτροπή Αναπτυξιακή Βοήθεια που θα γίνει στο Παρίσι 30 και 31 Οκτωβρίου. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι για αυτή τη συνεδρίαση τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου. Ο πρώτο είναι να εγκριθεί μια νέα εντολή για την Επιτροπή Αναπτυξιακή Βοήθεια που να συνάδει περισσότερο με τι αλλαγέ ε, στο διεθνέ πλαίσιο και ιδιαίτερα την ε, ατζέντα του 2030 και την ε, ατζέντα δράση τη Αντίσα Μπέμπα. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ξεκίνησε το 2012 για τον εξυγχρονισμό της ΝΤΑΚ ώστε να είναι κατάλληλη για την αναπτυξιακή συνεργασία του σήμερα. Στη διάρκεια αυτή τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου πρέπει να ληφθούν τέσσερι βασικέ αποφάσει. Πρώτον, η ανανέωση τη εντολή τη ΔΑΚ και του στρατηγικού οράματο. Δεύτερον, να πω ότι αυτό είναι απλώ μια εξέλιξη και όχι επαναστατική ε, δήλωση της ΔΑΚ. Κυρίω θα καθορίζει πρότυπα, θα ε, προωθεί την ε, ε, εκπαιδευτική διαδικασία και θα καθαρίζει και τα μέτρα στην αναπτυξιακή συνεργασία και υπάρχει ένα όραμα το οποίο περιλαμβάνει έξι διαφορετικά πράγματα, κινητοποίηση πόρων, εκπαίδευση, καινοτομία, επιρροή και αποτελεσματικότητα σε εσωτερικό επίπεδο. Το δεύτερο αφορά την έγκριση του μέσου επιλεξιμότητας του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μια συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το 2012 και είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή, ε, το 2014 ήταν συγγνώμη, σημαντική στιγμή, όταν υπήρχαν ε, τα ισοδύναμα μέτρα για τη χρηματοδότηση και τις δανειοδοτήσεις ε, σε ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να έχουμε ένα αντίστοιχο επίπεδο και για τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μια πρόταση αναχείρας και το βασικό στην πρόταση αυτή είναι μια μετάβαση από μια προσέγγιση ε, ροής μετρητών ε, σε ε, ισοδυναμία. Και αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί. Και το τρίτο είναι μια έγκριση κάποιων αρχών για την ε, συνδυασμένη χρηματοδότηση. Βλέπουμε ότι στην ατζέντα της Αντίσα Μπέμπα ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετέχει και ο ιδιωτικό τομέα ε, για να επιτύχουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και επομένω πρέπει να υπάρχουν και κάποια εργαλεία τα οποία κινητοποιούν ε, ιδιωτική χρηματοδότηση για να υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμό επιδοτήσεων και ε, δανειοδοτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορους φορείς, υπάρχουν κάποιες αρχές για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η συνδυασμένη χρηματοδότηση. Επισημαίνουν επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ευθαγραμμίσουμε και με τις αρχές αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για να είναι πολύ σημαντικά, για να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και ε, να έχουμε και μια προστιθέμενη αξία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να αντιμετωπίσουμε και τις αποτυχίες της αγοράς χωρίς να, να υπάρξουν ε, στρεβλώσεις της αγοράς. Θα υπάρξουν λοιπόν προτάσεις ε, και το τέταρτο σημείο είναι η έγκριση διευκρινήσεων για τη στατιστική οδηγία ε, και την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Δεν έχει αλλάξει η επιλοξιμότητα των δραστηριοτήτων, επομένως ο καθορισμός ε, παραμένει ο ίδιος. Αυτά τα οποία γίνονται τελευταία είναι η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται εκθέσεις από τα μέλη της ΔΑΚ για να υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας για την ερμηνεία του κώδικα. Και πάλι λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών, αυτής της ομάδας εργασίας θα υποβληθούν στην ΔΑΚ, στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Τώρα, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις εν εξελίξει στην ΔΑΚ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την θέση της ε, με όλες τις γενικές διευθύνσεις και ε, με μια ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία έχει κάτι να ρωτήσει. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να γίνει η διαλπούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Έχει γίνει κάτι τέτοιο ή προβλέπετε ότι θα γίνει. Η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών γίνεται σε διάφορες φάσεις αυτής της διαδικασίας και με στα πλαίσια της ΝΤΑΚ δηλαδή η ομάδα εργασίας για την χρηματοδότηση εμπλέκει και την κοινωνία των πολιτών. Άρα διαβουλευόμαστε με την κοινωνία των πολιτών σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ναι, η κοινωνία των πολιτών είναι ενήμερη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε την ημερήσιες διατάξει αυτών των ε, συναντήσεων, να ξέρουμε ποια είναι τα επόμενα θέματα και να μας πείτε, να διαβάζουμε και τι συνέβη. Δεν ξέρω κατά πόσο δημοσιοποιούνται όλα αυτά, αλλά να ξέρουμε τι συμβαίνει στον όσα. Δηλαδή ένα κατάλογο των συναντήσεων που προβλέπονται. Ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μακροχρόνια, αλλά και για την παρούσα, παρούσα περίπτωση μπορούμε να σας δώσουμε την ημερήσια διάταξη και υπάρχουν και έγγραφα αίθουσα. Δεν είναι δημοσιοποιημένα, αλλά μπορούμε να σας τα δώσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και ένα άλλο ερώτημα της Judith Sargent τίνι για την ε, ε, διαδικασία Κίμπερλι, αλλά στις 5 πρέπει να φύγουμε. Ε, λυπάμαι που προσήλθατε, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε αν η κυρία Σαρτζεντίνη δεν είναι εδώ. Θα το δούμε κατά την επόμενη συνάντηση έγκαιρα σε σχέση με τη διαδικασία Κίμπερλι και ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα όνομα το δικό μου ας πούμε για να δοθεί απάντηση. Ζητώ συγγνώμη από την Κομισιόν που προσήλθε. Λοιπόν, 18 διάφορα. Δεν μου έχει κοινοποιηθεί τίποτα. Στις 20 Νοεμβρίου στις 3 θα συναντηθούμε καθώς και στις 21, 9 με 12.30, 5 με 6.30 και έχουμε μία ακρόαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα περνάμε στην αίθουσα 2Q2 για το βραβείο Ζαχάροφ. Λυπάμαι που προσήλθε η Επιτροπή.